Νομίζω λοιπόν ότι φτάσαμε στις 3 και 20. Δεν φαίνεται να χρησιμοποιούμε όλοι τις ίδιες ζώνες ε, χρόνου. Λοιπόν, καταρχά σα ε, υιοθετήσουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν προτάσεις για αλλαγέ. Ευχαριστώ. Θα περάσω στις ανακοινώσεις. Έχω κάποιες. Πρώτον, Υπάρχουν ε, οι επόμενες συναντήσεις μας, την 4η Ιουλίου στο Στρασβούργο. Το βασικό θέμα θα είναι ανταλλαγή απόψεων με την Πολωνική Προεδρία των Οικονομικών τον Υπουργό, τον κύριο Σκόφσκι. Λοιπόν, στις 10 Ιουλίου έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Αλμούνια και τον Επίτροπο Σεμέτα επίσης Θυμίζω τις 31 ε, Αυγούστου, μετά τις διακοπές δηλαδή και το πρωί και το απόγευμα, έχουμε μια ολόκληρη μέρα δουλειάς, 31 Αυγούστου. Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτήν την συνεδρίαση, έχουμε πολλές εκθέσεις, θα γίνουν και δύο ψηφοφορίες εκείνη την ημέρα και μια ανταλλαγή απόψεων με τον Jean-Claude Crichet ως πρόεδρο της USRB. Κανονικά είχαμε πει να το κάνουμε στις 11 Ιουλίου, αλλά χρειάστηκε να αλλάξει η μέρα. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση και στην Ελλάδα και αλλού επιβάλλουν συνέχεια ε, περαιτέρω συναντήσεις και αλλαγές ημερομηνιών ανάλογα με τα γεγονότα. Τώρα για τον φάκελο των συναποφάσεων η Επιτροπή ΕΚΟΝ ψήφισε την έκθεση για το πρόγραμμα των εγγύησεων καταθέσεων. Ο διαπραγματευτής θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης, εφόσον πλέον το Συμβούλιο μπόρεσε να καταλήξει σε μια κοινή θέση. Η διαπραγματευτική εντολή θα καθοριστεί από την έκθεση της ΕΚΟΝ και η διαπραγματευτική ομάδα είναι ο πρόεδρος, ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές, ως συνήθως, εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Η διαδικασία λοιπόν θα συνεχιστεί. Ο εισηγητής μπορεί να πάρει και το λόγο αν θέλει, αλλά δεν το θέλει. Σάιμον. Σύντομα, μια παρατήρηση. Οι θέσει ε, διαφέρουν τόσο πολύ ώστε μπορούμε να πάμε κατευθείαν στη δεύτερη ανάγνωση, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε ούτω ή άλλω. Ε, ε, είναι τόσο πιεσμένο το χρονοδιάγραμμα που μόνο μία συνεδρία θα έχουμε πριν τι καλοκαιρινές διακοπέ και μετά από Σεπτέμβρη μπορούμε να περάσουμε στον τριμερή διάλογο. Okay. Um, then the Committee voted on the 6th of June. στις 6 Ιουνίου η Επιτροπή ΕΚΟΝ μίλησε για την αύξηση των μετοχών στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης. Εφόσον δεν υπάρχει άλλο είμαι εγώ η Θα ήθελα να σας πω ότι θα ζητήσω να υπάρξει μια συμφωνία σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διαδικασίες. Η ομάδα θα περιλαμβάνει εκτός από εμένα σαν εισηγήτρια και πρόεδρο του οι εισηγητέ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση γύρω από αυτό. Αυτή θα είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της έκθεσης μπορεί να γίνει και μέσω της γραπτής διαδικασίας. Σας είπα λοιπόν ότι η συνάντηση <coughs> με τον Τρισέ θα γίνει στις 31 Αυγούστου και όχι στις 11 Ιουλίου. Συγγνώμη σα ξαναλέω τα ίδια πράγματα. Εσείς θα γυρίσετε από τις διακοπές και θα ξεκινήσετε αμέσως δουλειά. σχετικά με τις ε, τεχνικές προϋποθέσεις για τις μεταφορές πιστώσεων η ψηφοφορία αναβάλλεται θα γίνει 11 και 12 Ιουλίου. Περνάμε τώρα στο σημείο 4 και το μέλλον του ΦΠΑ. Ο κύριος Κάζα έχει το λόγο. Κάζα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως καλωσορίζω την πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν. Το τωρινό σύστημα του ΦΠΑ δεν ταιριάζει στην εσωτερική αγορά. Το κόστος ε, συμμόρφωσης και το διοικητικό είναι πάρα πολύ υψηλό και βεβαίως το φέρουν ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι ευάλωτο σε απάτη, ειδικά όταν μιλάμε για συνοριακέ συναλλαγές όπου στη, έχουμε τη χειρότερη μορφή, την απάτη καρουσέλ που κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ στα κράτη-μέλη κάθε έτος. Τώρα είναι δύσκολο να βρούμε τι είναι το καλύτερο να κάνουμε και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Συναντήθηκα με εκπροσώπους μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων και ε, θα σας ε, αναφέρω τα βασικά μας συμπεράσματα. Ένα από τα θεμελιώδη σημεία που αναφέρονται στην έκθεσή μου είναι να αναγνωρίσουμε το status quo και να πάμε προς την κατεύθυνση του προορισμού όταν μιλάμε για τη φορολογία διασυνοριακού εμπορίου. Η θέση αυτή συμπεριλαμβάνει, έχει πάρα πολλούς ε, υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων ε, και η πράσινη βίβλος της Κομισιόν, όπου λέει πως ίσως η αρχή της προέλευσης να είναι καλύτερη για την εσωτερική αγορά. Οι απόπειρε των να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν αποτύχει. Η πολιτική βούληση δεν υπάρχει και άρα πρέπει να βρούμε μια κατάλληλη εναλλακτική. Ένα σύστημα που βασίζεται στην αρχή του προορισμού μπορώ να είναι αποτελεσματικό μόνο εάν υπάρχει μία υπηρεσία που να ασχολείται με τον ΦΠΑ. Η έκθεση υποστηρίζει αυτό το σχέδιο για τη σύσταση μίας υπηρεσίας αρμόδιας για τον ΦΠΑ μέχρι τον Ιανουάριο του 2015. Έτσι θα μειωθεί δραματικά το διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις και θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα διασυνοριακών συναλλαγών. Είναι ανησυχητικό πως ε, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχα, πολλοί ε, συνομιλητές μου παρατήρησαν πως προτιμούσαν να συναλλάσσονται με τρίτες χώρες παρά να ασχοληθούν με ε, ενδοκινοτικό εμπόριο στην υποτίθεται ενιαία αγορά, λόγω ακριβώς πολυπλοκότητας του συστήματος. Η κατάσταση αυτή βεβαίως είναι ανησυχητική και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Όσον αφορά τώρα τις επιλογές συλλογής του ΦΠΑ, είναι σαφές πως πρέπει να γίνει περισσότερη έρευνα για να δούμε τις ε, καλύτερες δυνατές επιλογές. Από τη συζήτηση και την ανάλυση που έκανα, θεωρώ πως ε, αυτό το οποίο αξίζει να μελετήσουμε περαιτέρω είναι ένας ε, συνδυασμός αποθήκευσης δεδομένων και δεδομένων ΦΠΑ, κάτι το οποίο βεβαίω σημαίνει επενδύσει σοβαρέ ε, σε υποδομές, γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και προτείνω περαιτέρω ανάλυση. Επίσης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε μια γενικότερη μείωση του κόστου συμμόρφωσης. Ε, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και οι οποίες δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα του συστήματος προτείνονται πολλές αλλαγές που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα χωρίς σοβαρές αλλαγές στο υπάρχον σύστημα. Η έκθεση ζητάει από την Κομισιόν να ε, υποβάλει ένα υπόδειγμα τιμολογίου το οποίο θα ε, είναι ουδέτερο γλωσσικά, δηλαδή να υπάρχει ένας πίνακας και θα ανταποκρίνεται σε κάποια εναρμονισμένα δεδομένα και δεν θα χρειάζεται άρα να υποχρεώνεται κανείς να μεταφράζει. Μεταξύ άλλων ε, συστάσεων προτείνεται να υπάρχει μείωση στη συχνότητα των ε, επιστροφών ε, ΦΠΑ οι αποδείξεις οι οποίες χρειάζονται για εξαίρεση από το ΦΠΑ να απλοποιηθούν, να χρησιμοποιηθούν λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσον αφορά υποβολή επιστροφών και να καταργηθούν ε, οι αναφορές ΦΠΑ ε, για ενδοκινοτικές συναλλαγές. Επίσης ε, θα πρέπει η Κομισιόν να ορίσει ποιες θα είναι οι μάξιμουμ υποχρεώσεις για ΦΠΑ. Οπότε αυτό σημαίνει πως τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν ήδη ένα αποτελεσματικό σύστημα δεν θα αυξήσουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στις επιχειρήσεις. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις θα έχουν την βεβαιότητα πως θα υπάρχει ένας οριστικός και εξαντλητικός κατάλογος υποχρεώσεων. Και θα πρέπει να παρακαλέσω τους συναδόλφους ε, βεβαίως και να συνεισφέρουν για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο κατάλογο. Οι επιχειρήσει ε, παλεύουν σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητα. Οπότε, ειδικά όσον αφορά ζητήματα τα οποία είναι μη επίμαχα, θα πρέπει να καταλήξουμε σε κανονισμούς και όχι σε οδηγίες για να αυξηθεί η πιθανότητα ενιαία ερμηνεία και εφαρμογής της νομοθεσίας περί ΦΠΑ. Αναμένω λοιπόν, είχαμε πάρα πολλές συνεισφορές και αναμένω βεβαίως συνεισφορά των συναδέλφων για να ακούσω τι θα πούν και οι σκιώδεις εισηγητέ για να αναζητήσουμε συμβαστικές λύσεις στις ερχόμενες εβδομάδες. Ελπίζω η συνεισφορά του Κοινοβουλίου, συζήτηση για το μέλλον του ΦΠΑ να βοηθήσει την Κομισιόν που σκοπεύει κατόπιν να προβεί σε μια στρατηγική ανακοίνωση για το μέλλον του ΦΠΑ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον συγητή για την προσέγγιση την οποία περιέγραψε, πάει σωστή κατεύθυνση. Ε, περιγράφει μια σημαντική επιλογή η έκθεση η οποία πρέπει να γίνει από την χώρα προέλευσης ή προορισμού για την συλλογή του ΦΠΑ, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία στα οποία διαφέρει η άποψή μας. Είναι ε, περίπλοκο το θέμα και ούτως ή άλλως θα υπάρχουν τέτοιες διαφορές. Για εμάς ε, κρίσιμη σημασία έχει να αντιμετωπίσουμε την απάτη του ΦΠΑ. Είμαστε υπέρ τη απλοποίηση οπωσδήποτε και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε κάποιες διοικητικές διατάξεις ε, που έχουν κάποια χρησιμότητα όσον αφορά την καταπολέμηση της ε, απάτης να μην καταργηθούν έτσι απλά. Ε, π.χ. η συχνότητα περί αναφορών για την επιστροφή ΦΠΑ, η τρίμηνη, είναι σημαντική για να ανοιχνευτεί η απάτη, αλλά έχει και θετικά αποτελέσματα και για την ε, οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων. Θα πρέπει δηλαδή να αποφύγουμε το να πληρώνουν μία φορά το έτος το, το ΦΠΑ, γιατί σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να συγκεντρώνουν μεγάλα ποσά ε, συμφωνώ με την ιδέα της μίας αρμόδιας ε, υπηρεσίας. Θα πρέπει να το δούμε αυτό πώς θα είναι συγκεκριμένα και βεβαίως πρέπει να έχουμε σαφείς ε, ορισμούς. Οπότε εγώ θα έλεγα να έχουμε την έννοια κράτους μέλους χρήσης αντί για χώρα έδραση εγκατάσταση της χώρας για να αποφύγουμε ε, κατασκευάσματα όπου κάποιες εταιρείε είναι εγκαταστημένες π.χ. Ε, στο Μονακό και στην πραγματικότητα δραστηριοποιούνται στο λιμάνι της Αμβέρσας ή στο λιμάνι του Αμβούργου ή κάπου αλλού. Αυτό είναι στην παράγραφο 8. Επίσης ε, το ότι ο ΦΠΑ είναι μέσω πολιτικής το ύψος ε, του ΦΠΑ π.χ. ότι σε κάποιες χώρες ε, φτάνει σε κάποια προϊόντα το 6% ε, π.χ. για βασικά προϊόντα διατροφής είναι μια επιλογή πολιτικής ή αλλού ξέρω εγώ χρησιμοποιείται για να επηρεάσει μια οικολογική συμπεριφορά. Αυτό το οποίο λέει η Κομισιόν τώρα να φύγουμε από την επιβάρυνση του κεφαλαίου και να πάμε περισσότερο προς το ΦΠΑ δεν μας βρίσκει σύμφωνους ε, ως ε, ομάδα. Εμείς είμαστε υπέρ ενός φόρου χρηματοοικονομικών συναλλαγών, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση τώρα. Εκεί που λέει ο εισηγητής για το να αφαιρείται και να υπάρχει πλήρης έκπτωση του ΦΠΑ σε ορισμένες περιπτώσεις και εδώ πέρα δεν συμφωνούμε. Όπως είπαμε είναι ένα μέσω πολιτικής ε, δεν είναι δυνατόν να εκπίπτει από παντού ο ΦΠΑ, ο ΦΠΑ με όταν μιλάμε για έξοδα εστιατορίου σε εταιρείε ή έξοδα παραστάσεως, δώρα δημοσίων σχέσεων και τέτοια δεν είναι δυνατόν. Αλλά πρέπει να δούμε και πάλι ποια θα είναι τα, τα αποτελέσματα για τους ενδιαφερόμενους. Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών να είμαστε ουδέτεροι στο ΦΠΑ. Γιατί να διακρίνουμε μεταξύ αεροπορικών μεταφορών και σιδηροδρόμων. Γιατί ο ένας πληρώνει, ο άλλος δεν πληρώνει ΦΠΑ. Πρέπει να δούμε λοιπόν την ε, διοικητική απλοποίηση στα ενδοκινοτικά πύχη στις θαλάσσιες μεταφορές είναι πάρα πολύ πολύπλοκα και θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει κάτι στην έκθεση, αλλά τέλος ε, να πω το εξής. Υπάρχουν κάποιες ε, δραστηριότητες ε, που απαλλάσσονται και για λόγους πολιτιστικούς κτλ. Αν ε, επιβάλλουμε εκεί πέρα ΦΠΑ σημαίνει πως θα έχουμε και περαιτέρω κόστος γιατί θα αρχίσουν να ασχολούνται με λογιστικά και να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες για αυτόν τον τομέα. Αυτά και βασίστηκα σε αυτά τα οποία έγραψε ο εισηγητής και νομίζω πως ε, πάνω σε αυτά θα καταθέσουμε και τροπολογίες, αναμένουμε τη συνεργασία ε, για να έχουμε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον κύριο Κάζα που έχει επιτελέσει πολύ αξιόλογο έργο σε ένα εξαιρετικά δύσκολο όπως όλοι γνωρίζουμε θέμα. Ξεκίνησε κάτι τέτοιο το 1954 στη Γαλλία και στη δική μου πατρίδα θεσμοθετήθηκε ο ΦΠΑ το 60-61 και μάλιστα τότε ο Υπουργός Οικονομικών είχε υποσχεθεί ότι θα, είναι, θα ανέρχεται σε 1,5 με 2% το πολύ και μάλιστα θα ισχύσει μόνο για μια μεταβατική περίοδο διετή. Και τώρα έχουμε φτάσει στο 25% ΦΠΑ. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα πρέπει πάντως κάποιες αρχές να τις λάβουμε υπόψη. Παρόλο που μπορεί στη τελική ανάλυση να μην θεωρήσουμε ότι υπάρχουν ε, αρχές. Η πράσινη βίβλος προβλέπει ε, μετάβαση από άμεση σε έμεση φορολογία. Για πολλές χώρες αυτή η μετατροπή θα σημαίνει μια μετατροπή στην χρηματοδότηση του συστήματος πρόνοιας, ή ευημερίας μάλλον, και αυτό θα δημιουργήσει τρομερά προβλήματα σε ορισμένες χώρες τουλάχιστον. Βέβαια, έχει νόημα να γίνει μια μετακύληση του φορολογικού άχθους, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολο αυτό. Άλλωστε εδώ δεν, έχουν, δεν ισχύει η διαδικασία συναπόφασης. Προτείνεται και μία σύγκληση των συντελεστών ΦΠΑ. Αναφέρονται τα ποσοστά 18 με 25% σύγκληση γύρω από εκείνα τα ποσοστά. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει αύξηση της φορολογίας. Όχι μόνο τη φορολογική βάση, αλλά και τους φόρους για τους ε, φορολογούμενους. Αναφέρθηκε το πρόβλημα τη χώρα προέλευσης και τη χώρα προορισμού. Ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση. Τη συζήτηση αυτή την είχαμε κάνει και επ' του γερμανικού συστήματος. Και σίγουρα θα αναχαιτιζόταν κάπως η φοροαπάτη και φοροαποφύγη. Ε, αν λάβουμε υπόψη την χώρα προέλευσης ε, και αυτή να πληρώνει αλλά τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Και αυτό διαπιστώνουν. Γι' αυτό ίσως έχει νόημα η μετάβαση προς τη χώρα προορισμού. Ε, βέβαια, η άλλη αρχή είναι το status quo και ίσως αυτή ήταν η πιο, θα ήταν η πιο σωστή. Ίσως έχετε δίκιο. Αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι εμένουμε στην αρχική πρόταση, στην χώρα προέλευσης και είναι καλύτερη και πιο αντικειμενική. Σε ό,τι αφορά τη γραφειοκρατία, το γραφειοκρατικό άχθος, σίγουρα στόχος μας είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και το διοικητικό άχθος, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι αλληλένοντα αυτά τα δύο θέματα της μείωσης γραφειοκρατίας και του γραφειοκρατικού διοικητικού άκθου. Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα έχουμε τεράστιες απάτες. Αυτό το φαινόμενο της ε, απάτης καρουσέλ, όπως λέγεται. Σε ό,τι αφορά τέτοιου απάτες, τελικά είναι μια τέρμονη διαδικασία και κανένας δεν πληρώνει σε τελική ανάλυση. Θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς εδώ. Τώρα, η εύρυθμη λειτουργία και αναφέρθηκε και το μοναπευθυντικό σύστημα, το One Stop Shop. Συμφωνώ φυσικά και ίσως χρειάζεται κάτι τέτοιο για να γίνει πιο λειτουργικό και αποδοτικό το σύστημα. Πάντως, έχω κάποιες τροπολογίες σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά τιμολόγια και την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Το αναφέρεται και εδώ και θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το σύστημα, γιατί πραγματικά σήμερα χρησιμοποιούμε μια πολύ παράδοξη και απερχιωμένη μέθοδο. Θα πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Εσωτερική αγορά. Ναι, αν δεν κάνω λάθο και ο Μάριο Μόντι αναφέρει το ΦΠΑ και το σύστημα αυτό στη δική του έκθεση. Γιατί να μην το αναφέρουμε και εμείς λοιπόν, να αναφερθούμε στην έκθεση Μόντι σε ό,τι αφορά την ε, ενίσχυση της ενίας αγοράς. Αναφερθήκατε και σε κάποιες εξαιρέσεις, σε απαλλαγές. Αν κατάλαβα καλά, είστε κατά των ε, εξαιρέσεων γιατί δημιουργούν πρόβλημα και στη εσωτερική αγορά. Συμφωνώ. Αλλά κάποιοι συνάδελφοι, όπως και εγώ, μπορούμε να συμφωνήσουμε με την αρχή, αλλά και εγώ και η χώρα μου χρειαζόμαστε κάποιες εξαιρέσεις. Εφόσον φυσικά δεν στρεβλώνουν την εσωτερική αγορά. Αναφέρθηκε ο τομέας της εστίασης, εστιατόρια. Μπορώ να σκεφτώ και άλλους κλάδους και μάλιστα όταν ήρθε ο Επίτροπος πριν από ένα μήνα, συζητήσαμε και το θέμα των εξαιρέσεων. Για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, για παράδειγμα. Και υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις. Τα ηλεκτρονικά βιβλία. in Κάποια απλά αγαθά. Δεν νομίζω ότι εξαιρέσει αυτών θα στρεβλώσουν την αγορά. Και παρόλο που έχουμε υψηλές αρχές, ε, μας ενώνει η πολυμορφία σε κάποιο βαθμό. Θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε κάποιο περιθώριο λιγμών και για εθνικές απαλλαγές ε, εξαιρέσεις. Νομίζω ότι και ελπίζω μάλλον ότι θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στην Επιτροπή μας και να δεχτείτε κι εσείς κύριε Σιγητά κάποιες εξαιρέσεις αν δεν είναι υπερβολικά αρνητικέ. Πάντως γενικώ συμφωνούμε με την προσέγγισή σας. Θα καταθέσω φυσικά κάποιες τροπολογίες. Εγώ ήδη έχω συντάξει ορισμένες τροπολογίες και γνωρίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι σκοπεύουν να καταθέσουν τροπολογίες. Πάντως πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ευρεία συμφωνία και σας ευχαριστώ για τη μέχρι τώρα προεργασία και το σχέδιο έκθεσης. Άλλος κανείς? Έλαβα ένα σημείωμα από το σχέδιο εισηγητή των μεταρρυθμιστών ε, και συντηρητικών που σας ευχαριστεί που λάβατε υπόψη πολλά από τα σχόλιά του, λυπάται για την απουσία του. Αντίστοιχο σημείωμα μου έστειλε και ο συντονιστή των μεταρρυθμιστών και συντηρητικών. Θα, το διαβιβάσω, θα διαβιβάσω τα δύο σημειώματα στον εισηγητή, παρόλο που επί τη ουσία δεν υπάρχει τίποτα καινούριο. Δεν χρειάζεται να στα διαβάσω. Και δεν βλέπω κανέναν εκπρόσωπο των Πρασίνων ή τη Δημοκρατία και Ελευθερία. Θέλει άλλο κανεί το λόγο για το θέμα αυτό. Ο κύριο Μοργάντη, δεν βλέπω καθαρά το όνομα από εδώ. Sì, coordinatore σαν συντονιστής της πολιτικής μου ομάδας έφτασα καθυστερημένος γιατί είχαμε προβλήματα με το αεροπλάνο. Το ψήφισμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί οι εθνικές προσπάθειες ακολουθούν διαφορετικές κατευθύνσεις και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, προκαλεί επιπλέον κόστος και σπατάλες, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις για την ομάδα μου είναι πάρα πολύ σημαντική η βοήθεια για τις μικρομεσαίες. Ζητώ λοιπόν οι διάφορες, τα διάφορα όρια για το ΦΠΑ να καθοριστεί σε ένα σωστό επίπεδο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν στη χώρα μου και στην υπόλοιπη Ευρώπη ένα πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό δίκτυο. Χρειάζεται βοήθεια λοιπόν για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί κανείς από τις μικρές επιχειρήσεις για να μπορέσει μετά να ολοκληρωθεί και να μεγαλώσει. Ας μπορέσουμε λοιπόν να καλύψουμε τις ανάγκες των μικρομεσαίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούντβιγκσον. θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα θέμα το οποίο ίσως σας φαίνεται λίγο συνηθισμένο σχετικά με τους κανόνες της ΦΠΑ. Ε, τους κανόνες που αφορούν το ΦΠΑ των φιλανθρωπικών οργανώσεων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Σε χώρες όπως η Σουηδία, Φιλανδία και άλλες χώρες υπήρξαν πολλά προβλήματα και ε, παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη εφαρμογή της ισχύουσας κοινοτικής νομοθεσίας. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει να δούμε το θέμα λεπτομερέστερα και ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε είναι στα πλαίσια της οδηγίας να καταστήσουμε ικανές τις χώρες μέλη να επιβάλλουν περισσότερες εξαιρέσεις για τον τομέα των, της κοινωνίας των πολιτών. Μακάρι να υπάρξει μια γενικότερη κοινωνική εξαίρεση από τους κανόνες επιβολής ΦΠΑ για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Βέβαια πρέπει να είναι κανείς πολύ επιφυλακτικός όταν επιβάλλει τέτοιου είδους εξαιρέσεις και ε, γι' αυτό απαιτείται να δώσουμε περισσότερα περιθώρια κίνηση στα κράτη-μέλη. Γενικότερα οι εξαιρέσει αυτές για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προωθούν αυτή την κοινωνία. Μια σωστά οργανωμένη κοινωνία των πολιτών είναι κάτι το θετικό για το σύνολο της κοινωνίας. Εγώ έχω εργαστεί πολύ από τα 14 χρόνια μου και εξακολουθώ να εργάζομαι στον τομέα αυτό. Έχω ασχοληθεί και με ένα ίδρυμα το οποίο φιλοξενεί 600 άτομα και επίσης σε μια μεγάλη περιφέρεια με πάρα πολύ μικρά αεροκατοικημένα νησιά, ασχοληθήκαμε και με τους πολύ νέους ε, κατοίκους της περιοχής και καταστήσα, τους καταστήσαμε ικανούς να γυμνάζονται, να αθλούνται και νομίζω ότι θα πρέπει να διευκολύνουμε αυτές τις προσπάθειες, αυτές τις δραστηριότητες. Δεν θα πρέπει να είναι τόσο δύσκολο να προβλεφθεί γραπτά η δυνατότητα χορήγησης αυτών των εξαιρέσεων από την επιβολή ΦΠΑ. Όταν μιλάμε για τέτοιες οργανώσεις, μιλάμε για οργανώσεις μικρής κλίμακας, δεν μιλάμε για εμπορικές δραστηριότητες. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν θα αυξήσει τα έσοδα των οργανώσεων αυτών, αλλά θα απλοποιήσει την γραφειοκρατία. Και γι' αυτό αυτοί οι οποίοι βοηθούν τον κόσμο στον τομέα τους θα διευκολυνθούν. Πρέπει λοιπόν να εξετάσετε πολύ πιο προσεκτικά το τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό και εγώ προσωπικά ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια σωστή ορθολογική λύση και να προωθήσουμε τις δραστηριότητες αυτές τις τόσο σημαντικές για την κοινωνία που βοηθά τους νέους ιδιαίτερα να βρουν τον δρόμο τους στην κοινωνία αργότερα. Ευχαριστώ, Ζων Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Κάζα. Να του πω ότι συμφωνώ φυσικά με τις προτάσεις του. Ακούγοντας τους μεν και τους δε, καταλήγω σε δύο-τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν θα πρέπει να γνωρίσουμε δύο πράγματα σχετικά με το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι ένας φόρος τον οποίο πληρώνει ο τελικός καταναλωτής. ο τελικός στόχος της συναλλαγής ή του προϊόντος. Ε, είναι ουδέτερο αυτό το φορολογικό σύστημα για τους ενδιάμεσους παραγωγούς και δεν ευνοεί ένα σύστημα διανοήσεις βάρος κάποιου άλλου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Δεύτερον, είναι ένας φόρος ευρωπαϊκού τύπου. Είναι ο μοναδικός πράγματι ευρωπαϊκός φόρος, στα πλαίσια του οποίου κάθε χώρα έχει αποδεχθεί θα έλεγα ένα υψηλό ποσοστό εναρμόνισης και στα πλαίσια των κανόνων του ΦΠΑ και της αναθεώρησής τους πιθανώς δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε το κριτήριο αυτό και θα πρέπει να προχωρήσουμε στη μεγαλύτερη δυνατή περαιτέρω εναρμόνιση για να μην πω για συνολική εναρμόνιση και έρχομαι εδώ σε αυτό που έλεγε ο Όλε Σμιντ ε, στις απάτες, γιατί το σύστημα αυτό περιλαμβάνει και υψηλά ποσοστά απατών, εφόσον έχουμε διαμεθοριακές δραστηριότητες μέσω του συστήματος καρουσέλ, γαϊτανακίου. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι ο φόρος αυτός είναι ένας ευρωπαϊκός φόρος, ένας έξυπνος φόρος, τον οποίο θα πρέπει να βελτιώσουμε. Μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις, απαλλαγές πιθανές κτλ. Θα πρέπει να είναι όσο λιγότερες δυνατές γίνεται. Δεν είναι ο ΦΥΠΙΑ ο τρόπος για να διευκολύνουμε τις ε, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Εξαιρετικός ο ρόλος τους. Αλλά δεν θα πρέπει με τη ΦΥΠΙΑ να τις βοηθήσουμε, αλλά με τις επιδοτήσεις, με τους φόρους που υπάρχουν στις χώρες εις βάρος των οργανώσεων αυτών και θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις οργανώσεις οι οποίες είναι σαφέστατα μη κερδοσκοπικές με συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους που περιέγραψε ο συνάδελφος και επίσης και την κακή χρήση αυτού του είδους των οργανώσεων και μιλάω για τη χώρα μου, τη Γαλλία, όπου τέτοιου είδους οργανώσεις χρησιμοποιούνται για κερδοσκοπικούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει είμαι βέβαιος ότι ο Νταβίντ Κάζα θα μας ε, δώσει μια εξαιρετική τελική έκθεση τη στιγμή που ξεκινάει μια ριζική αναθεώρηση του συστήματος ΦΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλους τους ομιλητές. Πρέπει να πάρω μια θήκη για τον Τέιβιτ, θέλεις να ακούσουμε την Κομισιόν. Ε. Κύριος έχετε το λόγο. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια πράσινη βίβλο ακριβώς ε, για να λάβει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις στα πλαίσια δημόσιων διαβουλεύσεων. Και τα τέσσερα πρωταρχικά σημεία που ανέφερε ο εισηγητής, το μελλοντικό σύστημα του ΦΠΑ, ε, επισήμαναν την ανάγκη ουδετερότητα αυτού του συστήματο, Σημαντικό θέμα η ουδετερότητα, γιατί ο τελικό καταναλωτή τελικά πληρώνει το ΦΠΑ. Και διαπιστώνουμε ότι στην πράξη πολλές φορές οι φορολογούμενοι ε, αντιμετωπίζουν αυτή την έλλειψη ουδετερότητας και αναλαμβάνουν ένα τμήμα του ΦΠΑ. Υπάρχει μια συνέπεια λοιπόν σε ό,τι αφορά τους διάφορους τομείς και μια διαφορά. Σε ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις ή τις παρεκκλήσεις ή τις απαλλαγές, Υπάρχει όντω ζήτημα. Μέχρι στιγμής και από την πρώτη οδηγία του 67 θέλησαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιδιώξουμε μια μεγαλύτερη εναρμόνιση. Ανακύπτει όμως εδώ το ερώτημα Θέλουμε ενίσχυση αυτής της εναρμόνισης ή μήπως θα πρέπει να αφήσουμε περισσότερη ελαστικότητα στα κράτη-μέλη, αρκεί βέβαια να μην υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού σε κοινοτικό επίπεδο. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύστημα της χώρας προέλευσης, ανακύπτει το ερώτημα κατά πόσο <clears throat> συντρέχουν οι προϋποθέσεις και αν υπάρχει πραγματικά γνήσια πολιτική βούλη στον κρατών μελών για να εφαρμόσουν ένα σύστημα χώρας προέλευσης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το σύστημα χώρας προέλευσης προτάθηκε από έξι κρατημέλη το 1967 και έχουν περάσει 44 χρόνια και μέσα 27 χώρες μέλη στην Ένωση. Οπότε ίσως θα πρέπει να συζητηθεί και πάλι το θέμα με όλα τα κράτη-μέλη. Ένα άλλο ζήτημα που ανακύπτει είναι ότι με την υιοθέτηση του πακέτου ΦΠΑ για το, τις παροχές υπηρεσιών ε, φαίνεται ότι ε, στρεφόμαστε προς ε, μια φορολογία στη χώρα κατανάλωσης και είναι λίγο δύσκολο να υπαναχωρήσουμε σχέση με αυτό. Σε ό,τι αφορά το μονοπευθυντικό σύστημα, το One Stop Shop, αυτό βέβαια θα διευκολύνει πολύ τους ε, διάφορους φορείς και χρήστες, παρόλο που η εφαρμογή πρακτική θα είναι κάπως δύσκολη. Το 2005 είχαμε μια πρώτη περιορισμένη στη εμβέλειες επιχείρηση. Τώρα να μειώσουμε τη, τις υποχρεώσεις ε, των φορολογουμένων, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη συλλογή του ΦΠΑ. Και θα πρέπει να βρούμε ε, μια ισορροπία μεταξύ του περιορισμού των περιττών υποχρεώσεων και της ανάγκης ε, εξασφάλισης της συλλογής του ΦΠΑ, συγκέντρωση ΦΠΑ. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση των ενδοκινητικών συναλλαγών, μερικοί μας είπαν ότι είναι πιο εύκολο ε, να κάνει κανείς εξαγωγές προς τρίτες χώρες παρά να έχει ενδοκινοτικές συναλλαγές. Και μας εκπλήσει αυτό, γιατί έχουμε εσωτερική αγορά. Θα πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε. Είναι φυσιολογικό να ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την ίσπραξη του ΦΠΑ, Στι περισσότερε χώρε ισχύει το ίδιο σύστημα με αυτό που ισχύει πριν από 40 χρόνια. Διαρωτόμαστε λοιπόν μήπω ήρθε η στιγμή να τροποποιήσουμε τον τρόπο συλλογή του ΦΠΑ χρησιμοποιώντα την τεχνολογική, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή. Και Αυτά φυσικά θα μπορούσε να γίνει μόνο μέσο πρόθεσμα. Μία άλλη σημαντική ερώτηση είναι η νομοθετική διαδικασία. Σε μια νομοθετική διαδικασία που προβλέπει ομοφωνία για τη φορολογία ε, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, ε, ο εισηγητής είναι υπέρ κανονισμού παρά οδηγίας. Βέβαια, η, η βάση για τη φορολογία είναι το άρθρο 113 της συνθήκης που δεν λέει τίποτα για τη νομική βάση ή για τα μέσα για το μέσο με τον οποίο θα επιδιωχθεί. Κάλιστα θα μπορούσε να υποβληθεί κανονισμό στη θέση τη οδηγία. Αλλά και εδώ περιορίζεται η ελαστικότητα που ζήτησαν ορισμένοι. Όλα αυτά τα ζητήματα μας προβλημάτισαν και στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου και σε αυτή τη φάση θέλουμε κάποιες ξεκάθαρες απαντήσεις. Βρισκόμαστε σε φάση δημόσιων διαβουλεύσεων. Μέχρι στιγμή έχουμε λάβει 1.700 συνεισφορέ, 8.000 περίπου σελίδε γράφων συγκεντρώσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπως είπε και ο συγητής πριν το τέλος του έτους θα υποβάλουμε ανακοίνωση με τους τομείς προτεραιότητας για το μέλλον στα θέματα ΦΠΑ. Αυτά προς το παρόν κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Thank you. Um, ευχαριστώ. Ο συγητής θέλει να δευτερολογήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ συνάδελφοι για τα καλά σας λόγια και την επικοδομητική συνεισφορά. Θα προσπαθήσω τώρα... Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα σχόλιά σας για αυτό το οποίο είπατε για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Να πω πως ε, ευθύς εξ αρχή συμφωνώ με το σκεπτικό αυτό και όσον αφορά αυτό το οποίο είπε ο κ. Σμιτ συναντήθηκαν πολλούς ε, ενδιαφερομένους ε, επ' αυτού, μεταξύ των οποίων και έναν ε, Σουηδό βουλευτή και είμαι διατεθειμένος να συζητήσω τη δυνατότητα να εισαχθεί αυτό το στοιχείο. Τώρα ο κύριος Λάμπερτ, ο οποίος οψιάζει σήμερα, όπως και ο κύριος Σμιτ, μου έστειλε Κάποιο ένα ενημερωτικό σημείωμα για τα ηλεκτρονικά βιβλία και την αρχή της ουδετερότητας. Όπως σημειώσατε, ε, υπάρχουν διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές στα ηλεκτρονικά από τα τυπωμένα βιβλία. Και παράγματι, όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 5, ε, υπάρχει αρχή πως παρόμοια αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση. Αντιλαμβάνομαι πως αυτό ίσως πρέπει να αναφερθεί πιο έντονα στην έκθεση και είμαι διατεθειμένος να συζητήσω τις προτάσεις σας για εναλλακτική διατύπωση. Όσον αφορά τις προτάσεις των, των σοσιαλδημοκρατών συναδέλφων, Ευχαριστώ. Ε, ακούω την στήριξή σας για την ε, αρχή προορισμού. Επίσης για την καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ συμφωνώ απολύτως και βεβαίως θα πρέπει να ενισχυθούν οι διατυπώσεις των σχετικών παραγράφων. Για το θέμα της απάτης επίσης συμφωνώ με τις ε, θέσεις που μου ανέφερε ο κύριος Λάμπερτς. Τώρα αναφέρατε και εξαιρέσεις. Δεν λέμε να μην φύγουν οι εξαιρέσει ε, εντελώς από την έκθεσή μου. Το καταλαβαίνω πως ε, κάποιες εξαιρέσει είναι πάρα πολύ σημαντικές για διάφορες χώρες. Οπότε αναμένω την συνεργασία μαζί σας για να δούμε την διατύπωση όσον αφορά και τις εξαιρέσεις. Αυτά είχα να πω για την ώρα κυρία Πρόεδρε. Αναμένω και τη συνεργασία με του συναδέλφου τι ερχόμενε εβδομάδε. Ευχαριστώ για την συνεισφορά και την υπομονή σα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάπου εδώ ήταν το πρόγραμμα. Λοιπόν, η 30 Ιουνίου είναι προθεσμία για τροπολογίες, εξέτασή του 31 Αυγούστου και σκοπεύουμε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας 19 Σεπτεμβρίου και πάλι στόχος είναι η δεύτερη ολομέλεια του Οκτωβρίου θα περάσουμε τώρα στην ακρόαση, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Βέρνερ Λάγκεν που δεν ήταν εδώ όταν ε, σας ενημέρωσα για τη συναπόφαση και τους τριμερείς διαλόγους και θα ήθελα νομίζω να μας πει ποιες είναι οι σκέψεις του για τη διαδικασία σχετικά με τον Εμμύρ. Ναι, πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα προχωρήσουμε στις 5 ε, του, του μηνός. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες, είτε να ολοκληρωθεί πλήρως η πρώτη ανάγνωση και να αναμένουμε το Συμβούλιο. Δεύτερη δυνατότητα να ολοκληρωθεί το νομοθετικό κείμενο, αλλά να μην κάνουμε τελική ψηφοφορία και να διαβουλευτούμε με το να διαπραγματευτούμε το Συμβούλιο. Και η τρίτη δυνατότητα είναι να ολοκληρώσουμε και να συνεννοηθούμε με το Συμβούλιο για μια συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση ή μια επίσης συνήθις διαδικασία. Σε όλες τις περιπτώσεις νομοθεσία απαιτεί να παρουσιάσει κάποιο αποτέλεσμα το Συμβούλιο. Δεν το έκανε αυτό επί Ουγγρικής Προεδρίας και υπήρχε μια συζήτηση προς ανατολισμού αλλά σύμφωνα με αυτά τα οποία είδα εγώ, δεν ξέρουμε πότε επί Πολωνικής ε, Προεδρίας ε, θα καταλήξουμε σε κάποια ενιαία στάση του Συμβουλίου. Και η ερώτησή μου είναι πώς θα προετοιμαστούμε. Έχουμε κάποιες τεχνικές τροπολογίες από πλευράς νομικής υπηρεσίας για πράξεις τα κτλ. Μετά έχουμε και τροπολογίες που αναμένουμε από κάποιου συναδέλφους και έχουμε τώρα τα, τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες. Εάν με ενημερώνουν σωστά θα είναι έτοιμα σε όλες τι γλώσσες ε, απόψε. Δεν ξέρω στο, στην αρχή ή στο τέλος συνεδρίασης, αλλά αυτό μας είχαν υποσχεθεί σήμερα. Και αυτό το οποίο πρέπει να αποφασιστεί τώρα είναι δύο πράγματα. Έχουμε αφενός ε, τις αλλαγές που προτείνει η νομική υπηρεσία και βεβαίως ένα θέμα είναι κρίσιμο εδώ πέρα, το εάν η ΕΣΜΑ είναι μία από τις αναγνωρισμένες αρχές, ε, αναφέρει δε η νομική υπηρεσία πως δεν αναφέρεται στη συνθήκη, παρά μόνο είναι μία ε, δευτερεύουσα αρχή, εδώ πέρα θέλω να στηρίξω εγώ τη θέση της ΕΣΜΑ και τα υπόλοιπα ζητήματα είναι τεχνικές αλλαγές, μπορεί να δεχτεί νομίζω η Επιτροπή. Και το δεύτερο ζήτημα είναι αν θα γίνει η τελική ψηφοφορία ή όχι. Εδώ πέρα θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις. Και στις δύο περιπτώσεις, χωρίς τελική ή με τελική ψηφοφορία, μία συμφωνία νωρί στην δεύτερη ανάγνωση είναι δυνατή μετά τι διακοπέ του καλοκαιριού εάν έχει συμφωνήσει βεβαίω σε μία θέση το Συμβούλιο και νομίζω μπορεί να γίνει αυτό και να ολοκληρώσουμε σχετικά γρήγορα. Οπότε είναι ανοιχτό το ζήτημα και θέλω να ακούσω τις, τις απόψεις σας για να διαμορφώσουμε και μία στάση. Γιατί υπάρχουν προθεσμίες και στόχος θα πρέπει να είναι τον Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου, να έχουμε τελειώσει έτσι ώστε να το αναλάβουν και οι λοιποί, η ΕΣΜΑ και οι λοιποί, για να κινηθεί η διαδικασία. Ζαν Πολ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημερίζομαι φυσικά την ανάλυση του Βέρνερ. Έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα και έχει πετύχει και μια μεγάλη πλειοψηφία στις θέσεις του στην Επιτροπή. Αυτό που έχει πάντως σημασία είναι στο θέμα αυτό να μην χάσουμε πια άλλο χρόνο και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που υπάρχουν για περαιτέρω ρυθμίσεις. Έχουμε δύο δυνατότητες. Είτε θα ψηφίσουμε επιμέρους ένα τμήμα τον Ιούλιο και θα αφήσουμε ανοιχτή την δυνατότητα για συμφωνία με το Συμβούλιο στην πρώτη ανάγνωση τις επόμενες εβδομάδες. Η λύση αυτή ξέρετε ότι έχει ήδη παρελθόν προηγούμενο και έχει ενδιαφέρον γιατί το Συμβούλιο πράγματι δεν έχει αποφασίσει ακόμα και το κείμενο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο με πλειοψηφία ισχυρή θα είναι ένα πρότυπο για να βρει λύση και το Συμβούλιο. Να σας θυμίσω εδώ τι είχε γίνει για τις υπηρεσίες πληρωμών, την οδηγία υπηρεσιών πληρωμών, όπου το Κοινοβούλιο είχε συμφωνήσει το Σεπτέμβριο του 2006, το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2007 και το κείμενο του Συμβουλίου εν πολλής αντικατόπτριζε τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Η δεύτερη λύση, για να μην σημειωθεί περαιτέρω καθυστέρηση, θα είναι να αναβληθεί η ψηφοφορία για όσες μέρες χρειάζεται, έτσι ώστε να συνταχθούν οι τροπολογίες τις οποίες αναφέρθηκε ο Βέρνερ και είναι υποσυζήτηση. Πάντως εγώ είμαι υπέρ μιας λύσης η οποία δεν αποκλείει αυτόματα την πρώτη ανάγνωση, ε, μόνο και μόνο για να κερδίσουμε κάποιους μήνες τελικά. Συνειδητοποιώ ότι οι υπόλοιποι σκιώδεις δεν είναι εδώ. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τους φιλελευθέρους και θα συμφωνήσω εν πολλής με αυτά τα οποία είπε ο Ζωαπόλ σχετικά με την κάλυψη των αναγκών και ότι θα είναι πιο εύκολο να καταλήξουμε σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης. Ίσως να έχουμε ανάγκη για αρκετούς τριμερείς διαλόγους. Ξέρω ότι ο Ζαν Πολ γενικά σκοπεύει να υπάρξουν στο θέμα αυτό πολύ, παρά να πιεστούμε στο εσωτερικό της δεύτερης ανάγνωσης. Λοιπόν, δεν έχουμε εκπρόσωπους των σοσιαλιστών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό την τελική απόφαση παρακαλώ να την πάρουμε στη συνάντηση της Δευτέρα στο Στρασβούργο, όταν θα έχουμε περαιτέρω διαβουλεύσεις ανάμεσά μας. Νόμιζα πάντως ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχετε την δυνατότητα να μας ενημερώσετε. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν που σας καθυστερώ όσους έχετε έρθει εδώ για την ακρόαση, για την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Θα ήθελα να ζητήσω επίσης συγγνώμη γιατί θα εγκαταλείψω την προεδρία της συνεδρίασης. Λυπάμαι που το κάνω αυτό γιατί το θέμα είναι προφανώς πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν θέματα στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης που θα έπρεπε να παρακολουθήσω, αλλά πρέπει να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σικλούνα για να συνεχίσει και να διευθύνει τη συνείδηση, την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Um, welcome to the public hearing on uh, the global economic governance. Um, as you know, we have a paper by. Λοιπόν, ξέρετε ότι ήδη έχουμε συζητήσει το θέμα που έχει παρουσιάσει ο κύριος Ρέκμαρκ. Θα ακούσουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων σήμερα. Σκοπεύαμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Πιέρ Ζαγέ, ο οποίος δεν έχει φτάσει όμως ακόμα και θα μιλήσει μετά από έναν-δυο άλλους ομιλητές. Στα πλαίσια λοιπόν της συγκυρίας, όπως είπε και η Πρόεδρος, το θέμα είναι πολύ επίκαιρο. Και περιμένουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας και τις απόψεις των ομιλητών. Θα μιλήσουμε για τις ε, εκκρεμότητες και ανισότητες ε, για τα θέματα των ευθυγραμμίσεων στον τομέα των ισοτιμιών. των τιμών των διαφόρων αγαθών και τις φούσκες στις τιμές αυτές. Στοιχεία ενημέρωσης λοιπόν για πιθανότητες μεταρρυθμίσεων σε όλους αυτούς τους τομείς, ιδιαίτερα στο Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. τις ε, προκλήσεις ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της ομάδας των 20 και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες αυτές τις αλλαγές και θα εμείνουμε λίγο και στα, ε, στους στόχους της Γαλλικής Προεδρίας της ομάδας των 20. Λοιπόν, ο κύριος Πιέρ Ζαγέ είναι Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας και θα μιλήσει εξ ονόματος της ομάδας των 20, αλλά δεν θα κάνει την εναρτήρια συνάντηση. Θα συνεχίσουμε με τους υπόλοιπους ομιλητές. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ροντόλφ Μπλαβή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ευρώπη, ειδικό σύμβουλος του Δέλτα Νιτάφ. Έχετε το λόγο και 7 λεπτά και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι ομιλητέ και στο τέλος εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις θα τις ακούσετε. Ευχαριστώ, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα εκ μέρου του Διεθνού Ομιζωτικού Ταμείου που είμαστε εδώ γιατί το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει. Είναι ένα ευρύτατο θέμα και για μας τα τελευταία χρόνια έχει καλύψει πολλά ζητήματα όπως την αναθεώρηση της εποπτείας, τροποποίησης ε, στις πολιτικές δανεισμού και ιδιαίτερα αναθεώρηση της διακυβέρνησης εντός του Διεθνούς Ταμείου. Ελπίζα ο πρόεδρος του G20 να σας δώσει μια γενικότερη επισκόπηση και εγώ να επικεντρωθώ σε ζητήματα του ΔΕΛΤΑ Αυτό θα κάνω λοιπόν και αν υπάρχουν ερωτήσει αργότερα πολύ ευχαριστώ να επανέλθω. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση εντός του Διεθνούς Ταμείου, Έχουμε πολλά επιτέγματα πρόσφατα και με αυτά θα ξεκινήσω πριν έρθω σε ευρύτερα ζητήματα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το ΔΕΛΤΑ και το προσωπικό του είναι υπόλογος κυβερνήσεις. Η δομή της διακυβέρνησής του απαρτίζεται από τρία σώματα. Το πρώτο είναι το Συμβούλιο των Διοικητών που συνεδριάζει άπαξ το χρόνο. Το δεύτερο σώμα είναι η Διεθνής ε, Νομισματική Επιτροπή Εποπτείας που, στην οποία συμμετέχουν ε, Υπουργοί Οικονομικών και Διοικητές Κεντρικών Τραπεζών όλων των χώρων μελών του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ και το Εκτελεστικό Συμβούλιο. Οι χώρες ε, εκπροσωπούνται στα διάφορα αυτά σώματα ανάλογα με το μερίδιό τους και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μερίδιο ε, για το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Τρεις είναι οι του, γιατί ε, προσδιορίζει τη συνεισφορά της κάθε χώρα στο κεφάλαιο του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Δεύτερος ρόλος είναι, καθορίζει το, το ποσό που μπορεί να δανειστεί κανείς από το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, αλλά και τις ψήφους που έχει στο εκτελεστικό συμβούλιο. Διοικητικό Συμβούλιο. Τα τελευταία δύο χρόνια το ΔΝΤΑΦ έχει επικεντρωθεί σε αυτό το θέμα των ποσοστώσεων και πέρυσι το Δεκέμβριο είχαμε μια σημαντική αλλαγή που έθεσε τέρμα σε μια αποτελμάτωση που είχαμε συναντήσει τελευταία δεκαετία ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσεις στο ΔΝΤΑΦ. Είχαμε πρόοδο σε δύο σημεία. Καταρχήν διπλασιάστηκε ε, το μέγεθος των μεριδίων σε 750 δισεκατομμύρια δολάρια και αυτό ήταν σημαντικό να ευθυγραμμιστούν οι πόροι του ΔΕΛΤΑ που μπορεί να δανείσει τα μέλη του με τις γενικές ε, ε, εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Επίσης είχαμε επανευθυγράμμιση των μεριδίων με, του, με τις ψήφους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η ευθυγράμμιση αυτή των μεριδίων ε, προήρθε από την δέσμευση των μελών του G20 να επαναθυγμίσουν το 5% των ε, ψήφων των ε, αναπτυσσόμενων χωρών προς τις χώρες που δεν εκπροσωπούνται ιδιαίτερα, όπως είναι οι αναφιόμενες οικονομίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με την απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου, το ΔΝΤ τήρησε αυτή την υποχρέωση και πάνω από 6% των ψήφων τις ε, μετέφερε από τις ανεπτυγμένες χώρες στις ε, ευρωπαϊκές χώρες και στις αναφιόμενες οικονομίες και αγορές. Τώρα, στην πράξη πώς λειτουργήσε το σύστημα. Ένα τρίτο των χωρών μελών του ΔΕΛΤΑ ε, βγαίνουν κερδισμένες από αυτή τη μεταφορά των μεριδίων. Και Έχουμε την Κίνα πια τον τρίτο μέτοχο στο ΔΕΛΤΑ και οι διαφορές μεταξύ των αναφιόμενων οικονομιών και των ανεπτυγμένων οικονομιών ε, μειώνεται όλο και περισσότερο. Το χάσμα γεφυρώνεται. Και βέβαια προσαρμογές αυτές οδήγησαν σε μια μείωση των δικαιωμάτων ψήφου για πολλές χώρες και αυτό επηρέασε κυρίως τις ευρωπαϊκές χώρες που έχανσαν 3,1% των ψήφων τους με τις τελευταίες αυτές μεταρρυθμίσεις του ΔΕΛΤΑ Αυτή ήταν η συμφωνία του Δεκεμβρίου. Βέβαια πρέπει να γίνουν και κάποιες ε, αλλαγές, να τεθεί σε ίσχυ καταρχήν η συμφωνία, κάτι που προϋποθέτει τη διπλασιασμό των, των μεριδίων, σε 70% την κύρωση από τις χώρες ε, μέλη και ε, την κύρωση για το 85% της μεταφοράς μεριδίων. Στην προηγούμενη μεταρρύθμιση που έγινε το 2008 χρειάστηκε Κάνουν δύο χρόνια για να εφαρμοστεί. Και προσπαθούμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη, να παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη του ΔΕΛΤΑ να κυρώσουν αυτές τις νέες μεταρρυθμίσεις. Για τις ευρωπαϊκές χώρες ποιες είναι οι συνέπειες. Μέχρι το 2012 θα πρέπει να αφήσουν δύο έδρες σε ευρωπαϊκές χώρες στο Διοικητικό Συμβούλιο προς όφελος των αναφιόμενων οικονομιών. αυτή η διαδικασία της εγκατάλειψης διαδρών από ευρωπαϊκές χώρες για ε, τις, για τις οικονομίες θα είναι ευκαιρία και για τις ε, ευρωπαϊκές χώρες να ξαναδούν πώς θα ε, κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί, πώς θα διαμορφώσουν πια την νέα τους παρουσία στο Δέλτα Νιτάφ. Και ίσως γίνει και μια αναθεώρηση των διαφόρων τρόπων των μεριδίων μέχρι το 2013, κάτι που ίσως ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία των αναφιόμενων οικονομιών στο Δέλτα Νιτάφ. Προσπαθήσαμε λοιπόν να αυξήσουμε στο Δέλτα Νιτάφ την εκπροσώπηση των αναφιόμενων αγορών και οικονομιών, αναπτυσσομένων χωρών και να γίνει καλύτερη ε, πανευθυγράμμιση και επαναπροσαρμογή με τη μετατροπή και με την μετατόπιση κάποιων μεριδίων. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό μέτρο για την νομιμοποίηση του ΔΝΤ. Φυσικά δεν είναι όλα μόνο αριθμητικά, δεν περιορίζονται σε νούμερα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που είναι σημαντικά και θα επικεντρωθώ σε τρία από αυτά. Ένα από τα μαθήματα που διδαχθήκαμε από την κρίση ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα φόρουμ οικονομικού συντονισμού πριν την κρίση. Μετά από αυτή τη διαπίστωση και μετά την κρίση κατατέθηκαν πολλές προτάσεις και από τον κύριο Τρέβορ Μάνουελ, από τον ε, ε, διαχειριστικό διευθυντή του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, που πρότεινε την ενεργοποίηση ενός ε, υπουργικού τέτοιου συμβουλίου με εκτελεστική όμως εξουσία εντός του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Ήταν ανάμεικτες οι απόψεις που ακούστηκαν. Ορισμένες, ορισμένοι παρατηρητές θεώρησαν ότι έτσι θα μειωθεί η εποπτεία σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι μόνιμο και τελικά προτιμήσαμε στις επιτροπές να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε τέτοιου είδους συζητήσεις και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις υπουργικές ε, δεσμεύσεις. Τώρα σε ό,τι φορά το γενικότερο ζήτημα της οικονομικής διακυβέρνησης και το σχετισμό G20 και ΔΝΤ, υπήρξαν προτάσεις ευθυγράμμισης της σύνθεσης του G20 με την ε, σύνθεση του ΔΝΤ. Για πολλούς και διάφορους λόγους, κυρίως γιατί πολλές χώρες αποκλείονται από το G20 και το σύστημα που προτάθηκε από την πρωτοβουλία Παλέρο Αγιάλ και αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής του ΔΕΛΤΑ είναι να, να ακουστεί περισσότερη φωνή και των αναπτυσσόμενων χωρών στη διακυβέρνηση, στα ζητήματα διακυβέρνησης. Ένα άλλο θέμα είναι το εκρεμές ζήτημα της διαδικασίας επιλογής για τον διαχειριστικό διευθυντή του ΔΕΛΤΑ Κάτι που είναι πολύ επίκαιρο αυτές τις μέρες. Με τη διαδικασία που ισχύει τώρα, που είναι η πιο ανοιχτή και διαφανής. Έχουμε δύο υποψηφίους για τη θέση του διευθυντού του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ που έχουν πολλά προσόντα. Ο ένας είναι από το Μεξικό, ο κύριος Κάρστενς, από αναφιόμενη δηλαδή οικονομία και η δεύτερη υποψήφια είναι η κυρία Λαγκάρτ, η Γαλλίδα Υπουργό Οικονομικών. Και το θέμα αυτό προχωρεί με τις δύο υποψηφιότητες. Βέβαια, το μείζον ζήτημα εδώ θα είναι πώς να χειριστούμε αυτό το θέμα και από τη σκοπιά του ΔΕΛΤΑ και από την πλευρά της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας ε, για ερωτήσεις ό,τι αφορά το διεθνές ε, σύστημα εποπτείας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, να πω κάποια πράγματα για τη σειρά των ομιλητών η οποία ανακατεύθηκε καθώς ήρθε και άλλος ένας συνάδελφος ο κύριο Ζέη. Θα του ζητήσω να μιλήσει στο τέλος. Και ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Χόκμαρκ που έπρεπε να είχε κάνει κανονικά την εισαγωγή. Αλλά θα μιλήσει πρώτος ε, όταν περάσουμε στις ερωταποκρίσεις. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο στον κύριο Αντρέ Σαπίρ, εταίρο του Ινστιτούτου Μπρούγκελ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να εμφανιστώ ενώπιον της Επιτροπής για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Να ξεκινήσω λέγοντας πως κατά την άποψή μου το σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης που έχει ε, πολλές ε, αδυναμίες, παρόλα αυτά ε, μας ε, έχει φανεί χρήσιμο και λειτουργήσε καλά στην ε, κρίση. Θα έλεγα πως το σύστημα αυτό είχε χάσει μεγάλο βαθμό νομοποίησης και θα μπορούσε να ανησυχεί κανεί για την ε, δυνατότητα να αντέξει ένα τόσο μεγάλο σοκ στην παγκόσμια οικονομία, αλλά νομίζω πως ε, αυτό δεν συνέβη. Το σύστημα λειτουργήσε ε, για να κάνει αυτό για το οποίο είχε σχεδιαστεί σε σχέση με τα διδάγματα του 1930 της εκείνης και αυτόν τον ρόλο έπαιξε ε, στην κρίση. Πράγματι, η G20 και ειδικά στη συνεδρίασή τους ε, του Λονδίνου τον Απρίλιο του 2009 ε, οπωσδήποτε αντέδρασαν στη, ισχυρά ως παγκόσμια κοινότητα και στην νομισματική πλευρά και στην πλευρά της βοήθειας δηλαδή μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας και λοιπόν διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Όσον αφορά δε το εμπόριο, ο προστατευτισμός μειώθηκε. Οπότε θα έλεγα πως αυτό το οποίο περιμέναμε εμείς ε, από το σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης ήταν ε, να μην κάνουμε τρομερά λάθη και να επιστρέψουμε στα 1930, το οποίο αποφεύχθηκε του του λεχθέντος είναι σαφές πως ήδη πριν από την κρίση το σύστημα το οποίο όπως σας είπα είχε δημιουργηθεί μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο με Bretton Woods, GATT που αργότερα έγινε POE και τα λοιπά το σύστημα αυτό ε, αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες. Αναφέρω δύο πράγματα. Το ένα είναι το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και το άλλο το σύστημα εμπορίου σαφώς ε, από την κατάρρευση του συστήματος του Bretton Woods ε, στις αρχές δεκαετίας του 1970 ε, βρισκόμασταν σε αυτό το οποίο πολλοί και εγώ περιγράψαμε ως ένα μη σύστημα και όσον αφορά το εμπόριο παρά το ότι ο ΠΟΕ λειτουργήσε κατά μία έννοια πολύ καλύτερα και έχουμε ένα παγκόσμιο σύστημα εμπορίου το γεγονός πως η γύρωση Ντόχα προχωράει ε, με πολύ αργούς ρυθμούς, να το πούμε έτσι, προφανώς μας δείχνει πως υπάρχουν πολλές ε, δυσκολίες. Τώρα, από πού προέρχονται αυτές οι δυσκολίες όσον αφορά το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και τον ΠΟΕ. Είναι συμπτώματα του ότι η παγκόσμια οικονομία εξελίχθηκε πάρα πολύ από όταν δημιουργήθηκε το σύστημα, όπως είπα, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια σημαντική εξέλιξη ήταν στην πλευρά των ΙΠΑ. Η οικονομία των ΙΠΑ και σε όρους οικονομικούς οπωσδήποτε από τη δεκαετία του 1980 δεν ε, είναι αυτό το οποίο ήταν όταν δημιουργήθηκαν αυτά τα θεσμικά όργανα. Ταυτόχρονα ε, οι ανερχόμενες οικονομίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι η Κίνα, παίζουν ένα ρόλο ο οποίος ήταν αδιανόητος πριν από 30 και 20 χρόνια. Και... Πάντα θέλω να θυμίζω ειδικά στους Ευρωπαίους πως ε, σχεδόν τυχαία όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ε, είχαμε το μικρότερο ποσοστό της Κίνας και της Ινδίας στον παγκόσμιο εμπόριο στην ιστορία και θα δούμε πως ο 20ος αιώνας ήταν μάλλον μια εξαίρεση ιστορικά μιλώντας. Οπότε τα θεσμικά όργανα τα οποία δημιουργήσαμε πριν από 60 χρόνια δημιουργήθηκαν σε, μια πολύ, ε, σε ένα πολύ ιδιαίτερο και συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι το ότι επιστρέφουν οι χώρες αυτές στο προσκήνιο και προφανώς ε, πρέπει να μεταρρυθμιστούν τα θεσμικά οργανά της παγκόσμιας διακυβέρνησης και ο ρόλος των χωρών αυτών πρέπει να αναγνωριστεί και νομίζω πως αυτό μόλις ακούσαμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να περάσουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Σκοπιά. Από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά υπάρχει σαφώς επιθυμία από πλευράς της Ευρώπης να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση ε, μόνο και μόνο γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια είναι μια πολυμερής κατασκευή και άρα θεωρεί θεσμικά όργανα παγκόσμιας διακυβέρνησης τα οποία είναι πολυμερή ε, τα βλέπει έτσι πολύ θετικά με την έννοια πως έχουν την ίδια φιλοσοφία ταυτόχρονα όπως είχα γράψει σε ένα βιβλίο του Ινστιτούτου Μπρούγκελ πριν από λίγα χρόνια, η Ευρώπη είναι μια κατακαιρματισμένη δύναμη με αδύναμη εσωτερική διακυβέρνηση σε πολλούς τομείς ε, εξωτερικής οικονομικής, εξωτερικής οικονομικής πολιτικής με κύρια εξαίρεση το διεθνές εμπόριο όπου μιλάει με μια φωνή στον ΠΟΕ. Επιπλέον, όπως ακούσαμε ε, από το Ταμείο, οι ευρωπαϊκές χώρες για ιστορικούς λόγους υπερεκπροσωπούνται στα θεσμικά όργανα του συστήματος Bretton Woods. Στα τελευταία δύο λεπτά που υποθέτω πως έχω ακόμα, να πω λίγα λόγια για μια έκθεση την οποία μόλις ολοκληρώσαμε με συναδέλφους τον Μπρούγκελ και το ΣΕΠΙ ε, για την Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ της Επιτροπής, όπου εξετάζουμε το μέλος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος εν μέρη από ευρωπαϊκή σκοπιά. Κοιτάμε τρία σενάρια του τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος τα επόμενα 10-20 χρόνια και βλέπουμε τρία σενάρια. Ένα το οποίο ονομάζουμε επισκευή και βελτίωση του υπαρχόντος συστήματος που σημαίνει σταδιακές μεταρρυθμίσεις Οπότε το σύστημα ως έχει με τον κυρίαρχο ρόλο του δολαρίου, αυτό το μη σύστημα, από το οποίο θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε κάποια βασικά προβλήματα, αλλά κάτω είναι επιστρέφουμε σε αυτό το σύστημα με οριακές μεταρρυθμίσεις. Ένα δεύτερο σενάριο είναι να πάμε προς ένα πολύ πολικό σύστημα το οποίο θα έχει χτιστεί γύρω από 2-3 νομίσματα κλειδί το δολάριο οπωσδήποτε και μετά πλην του δολαρίου το ευρώ και το κινέζικο γιουάν αλλά ένα... υπάρχουν και δυνατότητες πολυπολικών συστημάτων. Ένα διπολικό που δεν θα είναι δολάριο και ευρώ, αλλά διπολικό εννοώντας δολάριο και ερενμίνμπι, το κινέζικο νόμισμα, και ένα τρίπολιχο σύστημα ως εναλλακτική λύση που θα συμπεριλαμβάνει και το ευρώ. Τρίτο σενάριο, ένα πραγματικά πολυμερές σύστημα, δηλαδή κατά μία έννοια στο Bretton Woods, ακόμα και στις πρώτες μέρες του Bretton Woods θα έλεγα, με ένα πραγματικά πολυμερές διεθνές σύστημα με κεντρικό ρόλο για τα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα. Ένα πολυμερές, όχι πολυπολικό σύστημα θα το έλεγα. Τώρα, ποιο από αυτά τα σενάρια ε, είναι πιθανότερο. Όταν το σκεφτόμασταν αυτό, είδαμε το τι είναι πιθανό να γίνει και εκτός Ευρώπης και εντός Ευρώπης. Οπότε αυτό το οποίο πιστεύουμε είναι πως γενικά όταν βλέπουμε την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία πρέπει να δούμε τις εξελίξεις ε, στη ΣΥΠΑ, στην Κίνα, σε άλλα μέρη της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και τι συμβαίνει εντός της Ευρώπης, ποια είναι η δική μας δυνατότητα να οργανωθούμε. Η άποψή μας είναι, και εκεί πέρα προφανώς μιλάμε για την Ευρωζώνη, είναι πως ανάλογα με το πώς θα επιληθεί η τωρινή κρίση σε όρους οικονομικούς και διακυβέρνησης, το ευρώ στο δεύτερο σενάριο, το πολυπολικό, που δεν είναι οπωσδήποτε το πιο επιθυμητό ακόμα και από ευρωπαϊκή σκοπιά, το πολυπολικό θα ήταν ίσως το πιο επιθυμητό, αλλά και το πιο δύσκολο. Στο πολυπολικό λοιπόν αυτό σενάριο υπάρχει σαφής κίνδυνος το ευρώ να μην είναι ένας από τους πόλους. Εάν δεν καταφέρουμε να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας και από πλευρά οικονομικής και πολιτικής. Ευχαριστούμε κύριε Σαπίρ. Κιέρκεγκάρντ. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να είμαι μαζί σας σήμερα για να συζητήσουμε το θέμα της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Θα συγκεντρώσω τις σύντομες παρατηρήσεις μου στην ομάδα των 20, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στον ρόλο τον οποίο θα πρέπει να παίξει η Ευρώπη στους δύο αυτούς οργανισμούς. Η άνηση οικονομική ανάπτυξη συνεχίζεται με τις αναδυόμενες οικονομίες να αυξάνονται ε, και να εξελίσσονται τρεις φορές ταχύτερα από τις υπόλοιπες οικονομίες ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η οικονομική διακυβέρνηση είναι επίγον να τον δούμε. Οι αναδυόμενες οικονομίες αντιπροσωπεύουν το 50% της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και το μέγιστο ποσοστό της οικονομικής μελλοντική ανάπτυξης. Και παρόλα αυτά εξακολουθούν σε επίπεδο οικονομικής διακυβέρνησης να υποεκπροσωπούνται. Ο καθορισμός της ομάδας των 20 σαν τον βασικό φόρουμ για την διεθνή οικονομική συνεργασία μετά από την απόφαση της ομάδας αυτής στο Πίτσπουργκ δείχνει ότι υπάρχει μια κίνηση προς την συνολικότερη οικονομική διακυβέρνηση μετακινώντας την όμως από τις μεγάλες κυβερνήσεις οι οποίες την ελέγχουν σήμερα. Μετά από την αρχική αντίδραση στην κρίση του 2008 και 2009, η ικανότητα της ομάδας των 20 κατά τη διάρκεια μη ε, κρίσιμων περιόδων να ε, διακυβερνά την ε, διεθνή οικονομία είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα συζητήσιμο. Η διεύρυνση όμως της ε, ατζέντα της ομάδας των 20 είναι παράγοντες οι οποίοι δεν θα παίξουν και τόσο σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Η συνεχής απουσία μια ουσιαστική συνένεση στον τομέα της μακροπολι... μακροοικονομίας για την ομάδα των 20 και η έλλειψη ε, θα έλεγα επίσημων τυπικών δεσμεύσεων για τις κυβερνήσεις ε, να οδηγήσουν την οικονομική διακυβέρνηση σε συγκεκριμένα κοινά αποδεκτά επίπεδα, ε, θα έλεγα δεν μπορούν να στηρίξουν την επίτευξη των στόχων του ίδιου, της ίδιας της ομάδας των 20 για σταθερή και διαρκή ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν η ίδια η ουσία της ομάδας αυτής των 20 ίσως τελικά να περιορίζεται στα διάφορα διεθνή φόρα τα οποία συνεδριάζουν κατά καιρού ανάλογα με τις κρίσεις οι οποίες εμφανίζονται. Αναγνωρίζοντας αυτές τις ολοένα πιο ε, θα έλεγα επιταχυνόμενες αδυναμίες, βασικός μας στόχος θα, πρέπει να είναι να βελτιώσουμε τη λειτουργία των θεσμών της οικονομικής διακυβέρνησης. Η εμπειρογνωμοσύνη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ΟΑΣΕ και όπως επίσης και της, ε, Διεθνούς, της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι κάτι το αναμενόμενο. Η προώθηση λοιπόν της οικονομικής διακυβέρνησης στα πλαίσια της ομάδας των 20 θα πρέπει να οδηγήσει τους αρχηγούς των κοινευρωπαϊκών κυβερνήσεων να μην επιβαρύνουν την ομάδα των 20 με περιφερειακά θέματα σε σχέση με τον βασικό στόχο που είναι η επίτευξη μιας ισόρροπης και διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης. Δεύτερον, οι υπεύθυνοι για την οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βελτιώσουν τον ρόλο ειδικά του ΔΝΤ στα πλαίσια της οικονομικής ζωής και να συμπεριλάβουν και περαιτέρω πόρους για την αύξηση του ρόλου του στο ΔΝΤ και να βελτιώσουν τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των συστάσεων και των όρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία οικονομική χρηματοπιστωτική μάλλον κρίση επιβεβαίωσε τη μεγάλη σημασία που παίζει το ΔΝΤ η ενίσχυση λοιπόν του θεσμικού ρόλου και των διακυβερνητικών δομών του ΔΝΤ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωτικός και μια θα έλεγα ψύχρεμη αντιμετώπιση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει. Σαν συνεχώς μειούμενος διεθνός οικονομικός παράγων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εκτιμήσει τις δυνατότητες σφαιρικών παρεμβάσεων τις οποίες μπορεί να κάνει το ΔΝΤ και άλλοι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και να απομακρύνει θα έλεγα τις προκλήσεις οι οποίες είχαν καθοριστεί στα πλαίσια των πρώτων συναντριάσεων, συναντήσεων της ομάδας των 7 Νομίζω ότι μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της λειτουργίας του ΔΝΤ έπαιξε ένα πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν ο οποίος της αναλογούσε. Θα πρέπει λοιπόν τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τα επίπεδα διαχείρισης τα οποία έχει στο εσωτερικό του ΔΝΤ και στους άλλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς. Συνεπώς, είναι προς το συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης πριν από οτιδήποτε άλλο να προχωρήσει στην λεγόμενη μεταφορά Δυνατότητα ψήφου στο εσωτερικό του Δέλτα Νιτάφ προς τις αναδυόμενες οικονομίες και να μειωθεί η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δέλτα Θα πρέπει επίσης να βελτιωθεί η εξωτερική εικόνα και παρέμβαση του ευρώ και να βελτιωθεί επίσης και η εσωτερική οικονομική διακυβέρνηση του ευρώ και να υπάρξει ενιαία αντιπροσώπευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ΔΝΤ. Μια τέτοια συγκεντρωτική θα έλεγα ευρωπαϊκή παρουσία θα μπορέσει να καλύψει και τις εκτός ε, Eurogroup χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο θα την οδηγήσει βέβαια στο να χάσει δύο θέσεις στο ε, Διοικητικό Συμβούλιο του Δελτανιτά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία ε, ικανή και αντικειμενική για την επιλογή των ανωτέρων στελεχών του Νιτάφ και των άλλων οικονομικών οργανισμών χωρίς καμία αναφορά στην εθνικότητα του υποψηφίου ή στη γεωγραφική καταβολή και προέλευση ή δράση του συγκεκριμένου οργανισμού. Η Ευρώπη έχει να παίξει ένα ξεκάθαρο επικοδομητικό ρόλο προωθώντας επί της ουσίας και επί των ικανοτήτων τον υποψήφιό της ή την υποψήφιά της ε, για τη θέση του ε, Γενικού Γραμματέα του Δελτανιτά. Η βλαβερή πρακτική της περιφερειακής εναλλαγής που είναι θα έλεγα αποδεκτή σε επίπεδο διεθνών οργανισμών περιορισμένης πρακτικής όμως σημασία, δεν θα πρέπει να ισχύσει για οργανισμούς όπως το ΔΝΤ που έχουν κρίσιμους ρόλους να παίξουν στην διακυβέρνηση την οικονομική διεθνώς. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σας παρουσιάσω τις θέσεις μου σήμερα. Σας ευχαριστούμε κύριε Ακούσαμε τους ε, τρεις πρώτους ομιλητές μας. Ο πρώτος μας μίλησε για την κατάσταση των πραγμάτων ε, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο δεύτερος μας μίλησε για το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και το εμπορικό σύστημα και μας μίλησε για μερικές προτάσεις μεταρρύθμισής του και ο τρίτος ομιλητής μας μίλησε για το G20 και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός του G20 αλλά και εντός του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Θα ακούσουμε ναι. τώρα τον Πιέρ Ζαγέ που είναι ο Γενικός Διευθυντής ε, Διεθνών Σχέσεων και Έρευνας της ε, Τράπεζας της Γαλλίας και εκπροσωπεί εδώ την Προεδρία του G20. Εσείς δικαιούστε περισσότερο χρόνο, 10 λεπτά κύριε Ζαγιέ και περιμένουμε την ε, ομιλία σας. Η G20 είναι ένα διεθνές φόρουμ, σίγουρα, αλλά μια και η Γαλλία έχει την Προεδρία, θα αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία και θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, τα γαλλικά, αλλά μπορώ να απαντήσω μετά σε ερωτήσει και αγγλικά και γαλλικά. Θα ήθελα καταρχήν να σα ευχαριστήσω για την υποδοχή, τη θερμή υποδοχή και τη δυνατότητα που μου δίνετε να σα παρουσιάσω και τη Γαλλική Προεδρία στο G20 που βρίσκεται στα μέσα τη, γιατί έχουμε σε 4-5 μήνε τη διάσκεψη κορυφή των κανόν που θα μας δώσει κάποια αποτελέσματα, γιατί ακόμη βρισκόμαστε σε φάση προεργασίας. Και μάλιστα οι προεδρίες ακολουθούν μια συνέχεια. Το G20 δεν δημιουργήθηκε το 2008, παρόλο που το 2008 πήρε, απέκτησε νέα διάσταση. Το 1999 δημιουργήθηκε, μετά από πρωτοβουλία του G7, πρώτος πρόεδρος ήταν Καναδός, και η πρόταση, η ιδέα ήταν να γίνει καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών και των αναδειωμένων χωρών και οικονομιών. Και έτσι το 2008 είχαμε μια καινοτομία, το G20 έγινε πιο ορατό από πολιτική άποψη γιατί οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ε, συμμετείχαν σε αυτό το φόρουμ. Και όταν εξετάζουμε τις διαδοχικές ε, διασκέψεις κορυφής, τη της Washington του 2008 που ήταν μέσω της κρίσης, είτε τη διάσκεψη κορυφής του Λονδίνου που ήταν ε, μια διάσκεψη κορυφή που ασχολήθηκε με τα θέματα τη χρηματοπιστωτική ρύθμιση. Είχαμε τη διάσκεψη κορυφή του Πίτσμπεργκ που είχε ενδιαφέρον γιατί πραγματικά θεσμοθέτησε το G20 ως πρώτο φόρουμ για διεθνή οικονομική συνεργασία, όπως είχε αναφερθεί τότε. Στο Τορόντο ε, θεσπίστηκαν διάφορες υποχρεώσεις μακροοικονομικής πολιτικής και στη διάσκεψη κορυφής της υπό υποκορεατικής προεδρίας, Είχαμε το τέλος του, ενός κύκλου κατά κάποιο τρόπο, έγινε ένας απολογισμός διαφόρων θεμάτων και δόθηκαν και νέα σωθήσεις για άλλα. Η Γαλλική Προεδρία ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2010 και είχε ως προτεραιότητά της τέσσερα θέματα. Το πρώτο θέμα, συνεχίζοντας τις προηγούμενες προεδρίες, και κυρίως ε, της Κορέας ήταν να συνεχίσει τις εργασίες για μια βιώσιμη, ισχυρή και ισορροπημένη ανάπτυξη. Και νομίζω ότι υποτιμήσαμε κατά κάποιο τρόπο την ε, καινοτομία που συνιστά μια τέτοια πρόταση σε θέματα διεθνούς ε, μακροοικονομικής συνεργασίας. Υπάρχει βέβαια ένα τεχνοκρατικό σκέλος σε αυτή την προσπάθεια, αλλά για πρώτη φορά, κατά κάποιο τρόπο, οι χώρες για πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, θέτουν επιτάπητος διάφορες ε, υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που δεν είναι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά κυρίως μέσοπρόθεσμες και χρησιμοποιούν κάποια μέσα και διαρθρωτικής πολιτικής. Υπάρχει λοιπόν μια ισχυρή συνιστόσα δέσμευση, ε, ανάληψη υποχρέωση και αυτό είναι καινοτομία στο G20. Μια άλλη καινοτομία ε, ήταν το μια προσπάθεια που έγινε να κάνουμε και κάποιους μεσοπρόθεσμους μέσω, κάποιες μεσοπρόθεσμες προβλέψεις, να ταινίσουμε δηλαδή λίγο το μέλλον, περισσότερο όμως εξασφαλίζοντας μια συμπληρωματικότητα μεταξύ του ρόλου του G20 και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεν υπάρχει καμία προσπάθεια σφετερισμού υποκατάστασης, αλλά μια συμπληρωματικότητα. Μέχρι τις Κάνες θα έχουμε την ε, διαδικασία της αμοιβαία ε, αξιολόγησης που θα μας δώσει την ευκαιρία, θα δώσει την ευκαιρία στις περισσότερες χώρες του G20 και ιδιαίτερα στις 7 χώρες που εντοπίστηκαν ως ε, επιρρεπείς σε μεγαλύτερες ανισορροπίες, σε σοβαρότερες ανισορροπίες, να αναλάβουν κάποιες δεσμεύσεις και να πούν τι μέτρα προτίθενται να πάρουν προκειμένου να συμμετέχουν σε αυτό το συλλογικό σχέδιο για μια ισχυρότερη, βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη. Άλλο θέμα είναι το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Ένα ευρύτατο θέμα με πολλαπλές συνιστώσει που και αυτές είναι αλληλένδετες και συμπληρωματικές. Και μάλιστα συνεχίζονται στην Κορεατική Προεδρία, η Γαλλική Προεδρία επικεντρώσε στη συζήτηση στι διάφορε χρηματοπιστωτικέ δικλείδε ασφαλεία προκειμένου και να αποτραπούν κάποιες ε, ευνίδιες ε, διακοπές ιδιαίτερα σε οικονομίες που δεν έχουν τόσο ανεπτυγμένα κεφάλαια, να συνεχίσουν την ανάπτυξη σε καλές ηθίκες και να αποφευθούν κάποιες ρήξεις. Και φυσικά χρειάστηκε μια κινητοποίηση χρηματοπιστωτικών εργαλείων του ΔΕΛΤΑ αλλά και κινητοποίηση και άλλων μηχανισμών, γιατί στη διάρκεια της κρίσης είχαμε διμερή swap μεταξύ των κεντρικών τραπεζών και διάφορους άλλους μηχανισμούς. Η ιδέα λοιπόν ήταν να γίνει μια μεγαλύτερη, πιο σφαιρική, ανάλυση του ζητήματος της, της παγκόσμιας ρευστότητας προκειμένου να επιτρέψουμε στην, παγκόσμια οικονομία να έχει την απαραίτητη ρευστότητα και που απαιτείται όχι μόνο σε περίοδους κρίσης, αλλά γενικώ συνέχεια και ταυτόχρονα να αποφύγουμε spillover γιατί μερικές χώρες δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα μέσα οικονομικής πολιτικής τους. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και βρίσκεται στο πρόγραμμα της Γαλλικής Προεδρίας αυτή τη στιγμή. Τι είδους συμφωνίες μπορούμε να έχουμε σε διεθνές επίπεδο προκειμένου να υιοθετήσουμε ένα συλλογικό σύστημα για να μπορούμε να θεσπίζουμε κάποια μέτρα περιορισμού της ελευθερίας κεφαλαίων. Το θέμα αυτό βέβαια είναι μήλο της έριδας. Υπάρχουν μεγάλες διαμάχες μεταξύ των διαφόρων χωρών που έχουν μεταξύ χωρών που προσφέρουν ρευστότητα και αυτό που ζητούν. Να αποφευθούν αυτά τα spillover γιατί ορισμένες χώρες ε, που θέλουν να υιοθετήσουν κάποια μέτρα υιοθετούν νομισματικές πολιτικές που μερικές φορές ε, θεωρούν ότι έχουν ε, δυσμενή συνέπειες, ιδιαίτερα από τις ανεπτυγμένες χώρες. Είναι αρκετά επίμαχα αυτά τα θέματα, αλλά ελπίζουμε ότι θα προλαιώνουμε το έδαφος ώστε να καταλήξουμε στις κάνες σε μια συμφωνία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της δημοσιονομικής ρύθμισης. Ο βασικός στόχος της Γαλλικής Προεδρίας είναι καταρχήν να εφαρμόσει κάποιες ε, συλλογικές αποφάσεις και αποφεύγοντας τις ε, ε, ρυθμίσεις διαιτησίας και συνεχίζοντας τις προηγούμενες προεδρίες και της Κορέας και των προηγούμενων χωρών να θεσπίσει νέες υποχρεώσεις για το κεφάλαιο Βασιλεία 2 και 3 και να επεκτείνει σε όλο και περισσότερες χώρες αυτό το θέμα της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης που αρχικά προτάθηκε από το G20. Και τέλος για τις πρώτες ύλε. Το θέμα αυτό είναι αναφίβολα πολύ σημαντικό, αλλά και πάλι ιδιαίτερα επίμαχο, γιατί υπάρχουν εισαγωγή πρώτων υλών και εξαγωγή πρώτων υλών. Είναι πολύ μορφες οι αγορές πρώτων υλών, διαφορετική η ρυθμισή τους, υπάρχει μεγάλη ανομοιομορφία και ετερογένεια και δεν υπάρχει συμφωνία ούτε για τον τρόπο καλύτερη ρύθμιση αυτών των αγορών. Όλοι συμφωνούμε βέβαια ότι η μεταβλητότητα, η μεγάλη μεταβλητότητα αυτών των αγορών καλό θα ήταν να μειωθεί. Τέλος, τι πρόσφερε το G20 στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση. Ο, το Ιδρύμα Μπρίγκελ είπε ότι το G20 είναι μια ε, Διευθυντική Επιτροπή Οικονομικής Διακυβέρνησης. Κάτι που δείχνει ότι είναι ένα επιπλέον στοιχείο σε μια διαδικασία συντονισμού που, στην οποία συμμετείχαν και άλλες ε, οργανώσεις προηγουμένως και άλλοι θεσμοί. Επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια λογική συμπληρωματικότητα και όχι υποκατάσταση. Και εδώ θα ήθελα να τονίσω τον πολύ ενεργό ρόλο του Διεθνού Ομισματικού Ταμείου στη συζήτηση, ιδιαίτερα για τη μακροοικονομική πολιτική και το μακροοικονομικό συντονισμό στα πλαίσια του πλαισίου για μια βιώσιμη, ισορροπημένη και ισχυρή ανάπτυξη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει έναν αναδικατάστατο ρόλο και πραγματικά αποτελεί κινητήριο μοχλό και δίνει προτάσεις για τη λήψη μέτρων και την ποσοτικοποίηση των δημοσιονομικών αντικτύπων. Και προβλέπονται φυσικά και με τέτοια μέτρα από το G20 προτείνονται και από τον ΩΣΑ που επίσης διδραματεί σημαντικό ρόλο. Φυσικά η ζωή δεν είναι ένα ε, ήρεμο ποτάμι. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που ανακύπτουν και το G20 ήταν ένα θαυμάσιο εργαλείο σε καιρούς πολέμου. Ε, διαρωτόμαστε όμως αν θα είναι εξίσου καλός και αποτελεσματικός μηχανισμός και σε καιρούς ειρήνης. Και ίσως αυτή τη συζήτηση θα έρθουμε σε κάποια άλλη στιγμή. Υπάρχει και το θέμα της νομιμοποίησης που αναφέρθηκε από πολλούς. Το G20 αντιπροσωπεύει 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ και παρόλο που εκεί τυπικά δεν συμμετέχουν πολλές χώρες σημαντικών οικονομιών, παρόλα αυτά προσκαλούνται τακτικά στις συνεδρία του G20. Για παράδειγμα, η Αφρικανική Ένωση πολύ τακτικά συμμετέχει στις εργασίες του G20 και η ΑΣΕΑΝ. Άλλη πρόκληση είναι η λογοδοσία η ανάληψη ευθύνη. Το ότι είμαστε υπόλογοι ό,τι αφορά κάποιε δεσμεύσει που αναλαμβάνουμε. Και αυτή θα είναι πραγματική λιδία λήθο τη μακροοικονομική συνεργασία στα πλαίσια αυτού του πλαισίου που σας ανέφερα προηγουμένως. Καταρχήν οι χώρες σε καιρούς ειρήνης θα τηρήσουν αυτές τις υποχρεώσεις ε, προκειμένου να κινητοποιήσουν κάποιους ε, μηχανισμούς και εργαλεία για κυρίαρχη οικονομική πολιτική και να τη θέσουν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Και μπορούμε να έχουμε μία, έναν λεπτομεριακό απολογισμό του αποτελέσματος από την εφαρμογή τέτοιων μέτρων. Και υπάρχει και η πρόκληση της εξασφάλισης μιας συνέχειας. Το σύστημα της Τρόικας με τις α, τρεις προεδρίες είναι αποτελεσματικό, γιατί η συνεργασία δεν είναι πάντα εύκολη. Χρειάζεται μια μόνιμη συνεργασία. Ούτε για αυτό το θέμα υπάρχει συνένεση. Δεν πιστεύω ότι μια μόνιμη γραμματεία θα ε, πρόσθεται περισσότερη διαφάνεια σε μια ιδιαίτερα περίπλοκη τους ή οργάνωση με πάρα πολλές συνεδριάσεις, φόρα και ούτω καθεξής. Αλλά και αυτό το θέμα έχει τεθεί επιτάπητο κατά πόσο είναι αναγκαία και μία μόνιμη γραμματεία. Αυτά και περιμένω τι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ κύριε Ζωγέ. Θέσατε πάρα πολλά θέματα τα οποία ο κύριο Χερκμαρκ θα λάβει υπόψη του στα πλαίσια της ε, θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα λάβουν υπόψη τους επίσης και οι σκιώδεις εισηγητές. Ζητώ συγγνώμη κύριε Χόκμαρκ που δεν σας έδωσα το χρόνο να θέσετε το θέμα εισαγωγικά. Τώρα όμως αφού ακούσαμε τους ομιλητές θα έχετε την δυνατότητα πλέον να παρουσιάσετε μια ευρύτερη εικόνα του θέματος σαν εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι πράγματι τεράστιο. το βασικό που μπορεί να πει κανείς και το οποίο ανέφεραν όλοι οι ομιλητές είναι οι λεγόμενες αναδυόμενες οικονομίες. Εάν ήταν μόνο αναδυόμενες τότε το μέγεθος των προκλήσεων θα ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που είναι σήμερα. Το θέμα δεν είναι ότι αναδύονται, αλλά ότι αναδύθησαν. Είναι μια πραγματικότητα πλέον οι οικονομίες αυτές και νομίζω ότι όταν λέμε αναδυόμενες αυτό δείχνει το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Ε, είμαστε ο λίγο στραμμένοι στο παρελθόν. Δεν αναδύονται τώρα. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε με τέτοιο λαθασμένο τρόπο την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι έχουμε ε, φτάσει σε ένα εντελώς διαφορετικό διεθνές επίπεδο ισορροπίας σήμερα. Και οι οικονομίες αυτές μόνο αναδυόμενες δεν είναι. Εάν ήταν, η παγκόσμια οικονομία θα βρισκόταν στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν στο παρελθόν με πρωτοκαθεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δυτικής Ευρώπης. Και αν συνέχιζαν να αναδύονται, τότε θα είχαμε τις δυσκολίες που γνωρίσαμε στις ε, χρηματαγορές, αλλά δεν θα είχαμε την παγκόσμια, θα έλεγα, αλλαγή την οποία βιώνουμε τώρα και οι οικονομίες μας δεν θα ήταν τόσο θα έλεγα στενά διασυνδεδεμένες. Αλλά έχουν αναδυθεί πλέον οι οικονομίες αυτές και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο την αρχιτεκτονική των διεθνών οικονομικών οργανισμών. Δεν λειτουργούμε πλέον τόσο σε επίπεδο της ομάδας 7. Πολλοί αναφερθήκατε στην ομάδα 7, ομάδα 8, ακόμα και ομάδα των 10 που ήταν ένα στάδιο στην προσπάθεια αυτή της ε, απόπειρας ε, να δημιουργηθεί μια οικονομική διακυβέρνηση. Και το θέμα της Ελλάδας τώρα αντιμετωπίζεται όμως στα πλαίσια της ομάδας των 20. Αυτό δείχνει ότι η σημασία της οικονομικής διακυβέρνησης της διεθνούς έχει αυξηθεί ήταν σημαντικό θέμα και την εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Πολιτείε ήταν, όπως είπα, στην πρώτη γραμμή. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν υπάρχει πλέον μια κοινή πολιτική αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως το παρελθόν ίσως. Να σταθώ τώρα σε ένα βασικό πρόβλημα. Πόσοι οικονομική παγκόσμια διακυβέρνηση επιθυμούμε και πόσοι χρειαζόμεθα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το σταθμίσουμε. Αν προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όσο περισσότερη οικονομική διακυβέρνηση μπορούμε, τότε ο κίνδυνος αποτυχίας είναι πολύ μεγάλος γιατί θα έχουμε βάλει πολύ υψηλούς στόχους. Έχει σημασία λοιπόν να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στο τι είναι ουσιώδες και στο τι είναι επιτεύξιμο σε διεθνές επίπεδο και ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί τομείς με τους οποίους θα πρέπει να ασχοληθεί η διεθνής οικονομική διακυβέρνηση. Και φυσικά το θέμα των διεθνών ανισοτήτων ή ανισορροπιών αν θέλετε είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Η απάντηση σε αυτά τα προβλήματα εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο περιγράφονται τα ίδια τα προβλήματα. γιατί προσπαθούμε μερικές φορές να σχεδιάσουμε μια τέλεια σε εισαγωγικά διεθνή αρχιτεκτονική, αλλά ξεχνάμε να αντιμετωπίσουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα. Και υπάρχει εδώ και το θέμα του ρόλου των νομισμάτων, πράγματι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο και να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε νομίσματα όπως το νόμισμα της Κίνας. Είναι μετατρέψιμα βέβαια τα νομίσματα αυτά θεωρητικά, αλλά αν ήταν και επί της ουσίας τότε θα λύναμε κάποια σημαντικά ποσοστά των διεθνών αυτών ανισορροπιών. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, πολύ συχνά ξεχνάμε ότι όταν συζητάμε όλες, αυτούς τους, ε, όλες αυτές τις δομές της οικονομικής παγκόσμιας διακυβέρνησης, ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουμε να κάνουμε με πολυδιασπασμένη οικονομική πραγματικότητα σήμερα και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει την μέγιστη δυνατή επιρροή ε, στην κατάσταση. Εδώ θα ήθελα να ακούσω περισσότερα στοιχεία από τους φιλοξενουμένους μας σήμερα. Η ομάδα των 20 είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα θετικό βήμα θα έλεγα που ανταποκρίνεται και στις επιθυμίες του Κοινοβουλίου αλλά δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένας δημοκρατικός θεσμός, ένας διαφανής θεσμός, ένας θεσμός άμεσα αναγνωρίσιμος. Ο καθηγητής Σαπίρ αλλά και άλλοι είπανε ότι η ομάδα των 20 έκανε καλά πράγματα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αλλά βέβαια εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Έκανε θετικά πράγματα έτσι ώστε να μην επιδεινωθεί η κρίση αλλά ταυτόχρονα είδαμε ότι το σύστημα δεν μας έδωσε μια νέα λύση σε σχέση με τη μελλοντική υποδομή την οποία χρειαζόμαστε, γιατί θα πρέπει να αποφεύγουμε τέτοια λάθη και πρέπει να έχουμε τη δομή για να το κάνουμε αυτό και αυτό έχει σχέση και με τον ρόλο της ανταπροσωπευτικότητας αυτής της δομής. Θα ήθελα λοιπόν τις απόψεις των συναδέλφων για την σωστή αποκατάσταση της ισορροπίας ανάμεσα στην υπάρχουσα δομή του ΔΝΤ και την ομάδα των 20. Γιατί έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα, δεν χρειάζεται να επαναφεύρουμε τον τροχό, εφόσον έχουμε το ΔΝΤ και τον καθολικό χαρακτήρα και τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της ομάδας των 20, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα αυτά στα πλαίσια μιας νέας διαφανούς δομής, στο εσωτερικό της οποίας η ομάδα των 20 θα έχει καθοριστικό ρόλο. Μια ομάδα η οποία όμως δεν θα είναι μόνο πολιτικά σημαντική, αλλά θα είναι και πολιτικά υπόλογη. Ευχαριστώ κύριε Χακμάρκ. Θέσατε πάρα πολλά θέματα. Δεν ξέρω αν θα τα καλύψουν και οι υπόλοιποι βουλευτές που θα θέσουν ερωτήσεις. Σε αυτή τη φάση θα δώσω από δύο λεπτά στον κάθε ένα από τους ομιλητές για να δώσουν απαντήσεις σε κάποια από τα σημεία στα οποία, τα οποία τους έκαναν μεγαλύτερη εντύπωση από κάποια άλλα. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για το ζήτημα του ποιες είναι οι βασικότερες ανισορροπίες. Σαφώς δεν μειώθηκαν αλλά αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης οι παγκόσμιες ανισορροπίες και η G20 στην ε, συνάντηση του Φεβρουαρίου του 2011 σε επίπεδο υπουργών και διοικητών ε, βρήκαν ε, κάποιους δίκτες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουμε το ποιες είναι οι ανισορροπίες ε, που θα πρέπει να παρακολουθούμε και μιλάμε για δημόσιο έλλειμμα και χρέος, δημόσιες αποταμιεύσεις και χρέος και εξωτερικές ανισορροπίες. Και βεβαίως κάποιες χώρες, η Κίνα κυρίως, ε, δεν ήθελε να χρησιμοποιηθεί ο όρος ε, ανισορροπίες ε, τρέχουσων συναλλαγών, γι' αυτό μιλήσαμε για εξωτερικές ανισορροπίες, εννοώντας βεβαίως ε, το εμπόριο και τις ροές. Αλλά σαφώς δεν έχει τελειώσει η υπόθεση. Αυτή τη στιγμή έχουμε βρει αυτά τα πράγματα, γιατί δεν έχει τελειώσει η ιστορία με τις ε, ανισορροπίες. Ε, αν δούμε συγκεκριμένες χώρες όπως την Ινδία, σαφώς το πρόβλημα της Ινδίας είναι η έλλειψη υποδομών που βεβαίως ε, θα μειώσει τις δυνατότητες της. Στην περίπτωση της Κίνας το βασικό πρόβλημα είναι όπως σας είπα, η ισορροπία αυτή, αλλά στην πλευρά της Ευρωζώνης υπάρχει σε, κάποια περίπτωση, σε κάποιες περιπτώσεις μελών ε, χαμηλή παραγωγικότητα, στην Ιαπωνία πολύ υψηλό δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ τα λοιπά. Οπότε όλοι αυτοί οι δείκτες λαμβάνονται υπόψη. Και βεβαίως ε, δεν είναι μόνο κάτι το βραχυπρόθεσμο, αλλά θα πρέπει και να εμβαθύνουμε την ε, υπόθεση αυτή, να λάβουμε υπόψη είναι άλλες μεταβλητές ε, που υπάρχουν μέσω μακροπρόθεσμα για να υπάρξουν και κάποια μέτρα. Τώρα για το θέμα του τι θα μπορούσε να γίνει και ποια είναι η προσθέμενη αξία των g σε σχέση με το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Υπήρχε βεβαίω και η Σύνοδος του Άσιγκτον το 2008 που μας δίνει ένα παράδειγμα του πώς έχουμε ένα φόρουμ το οποίο το χρειαζόμαστε γιατί αντιδρά αλλά και δρά προληπτικά και συνεδριάζει εντός λίγων ημερών και λαμβάνει κάποιες αποφάσεις για να κινητοποιηθεί όχι μόνο το ΔΝΤ αλλά και το Ευρωπαϊκό ε, Φόρουμ Συστημικής ε, σταθερότητα για να λάβει τέτοιε αποφάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπλεβί. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τις ερωτήσεις που είναι αλληλένδετες σε δύο λεπτά. Αλλά το ευρύτερο ερώτημα του τι μπορούμε να κερδίσουμε, να βγάλουμε από την παγκόσμια διακυβέρνηση, μπορούμε παραδείγματος χάρη να δούμε το ζήτημα αυτό του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος που είναι στην ημερήσια διάταξη της Γαλλικής Προεδρίας και σχετίζεται με το εάν ε, βρίσκουμε ξανά τον τροχό με αυτά τα οποία έχουν γίνει στο Δονητού. Βασικό πρόβλημα του Δονητού ήταν η εμπλοκή των Υπουργών. Και βεβαίως το ζήτημα αυτό του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος και των παραδοτέων, θα έλεγα, των στόχων του Δουνουτού, βλέπουμε πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσπαθεί να αποκτήσει έτσι περισσότερο λόγο εδώ πέρα. Υπάρχουν λοιπόν τέσσερα θεμελιώδη προβλήματα που υπάρχουν στο Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Το ένα είναι η απουσία ενός παγκόσμιου μηχανισμού προσαρμογών στις παγκόσμιες ανισορροπίες και από πλευράς λοιπόν παραδοτέων πηγαίνουμε, ε, προχωράμε στο μέλλον με τις εκθέσεις αυτές ε, των ε, επιπτώσεων, όπως ζήτησαν και οι G20. Επίσης δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο αντιμετώπισης των ροών κεφαλαίου και το ανέφερε ο κύριος Ζαγέ, αλλά έχουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για ένα καλύτερο πλαίσιο πολιτικής. Η κρίση επίσης ε, τόνισε το ότι δεν υπήρχε ένα σαφής μηχανισμός παροχής ρευστότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και εδώ πέρα πάλι είδαμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να υπάρχει ένας μηχανισμός θα έλεγα ασφαλιστικού τύπου για να υπάρχει μια γραμμή πίστοσης και πάμε προς αυτή η κατεύθυνση. Τέλος, για το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα κάτι σχετικό με τα νομίσματα. Πηγαίνουμε, αν πηγαίνουμε σε ένα πολυπολικό σύστημα και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μετάβαση. Και εδώ πέρα βεβαίω τίθεται το ζήτημα των ειδικών τραφικών δικαιωμάτων και πώς μπορούν να διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση. Σε όλα αυτά λοιπόν τα σημεία νομίζω πως ο κύριος Ζαγιέ είπε πως το το συμπληρώνει τους G20 και πράγματι αυτό συμβαίνει, αλλά όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, η πρόκληση τώρα για την ομάδα των 20 είναι να αποδείξουν πως μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και σε καιρούς μη κρίσης και όλοι αυτοί οι στόχοι πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κύριος Σαπίρ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με τον ε, προηγούμενο μελητή για να διακρίνουμε ε, τους G20 σε καιρούς κρίσης και σε πιο κανονικούς καιρούς. Σας είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους G20 να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα σε καιρούς ε, ήρεμους και σε καιρούς κρίσης. δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Οπότε, τι είναι αυτό το οποίο εγώ βρίσκω παρόλα αυτά θετικό για τους G20. Θα θέλαμε οι G20 ή κάτι τέτοιο, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπάρχει και το πρόβλημα το πρόβλημα της συνομοποίησης που έχει, γιατί οπωσδήποτε η G20 δεν είναι G7, G8, οι οποίοι G7, G8 ήταν ηταν ε, εκτο πραγματικότητας ε, προκρίση. Εγώ που είμαι παντρεμένο με μία ινδί, δηλαδή δεν μπορούσα να ανεχθώ τους G7, G8, να φέρνουν τον Πρωθυπουργό της Κίνας και της Ινδίας. Δηλαδή τι αλαζονία είναι αυτή. Σε τι κόσμο νομίζουμε ότι ζούμε τελείως μη ρεαλιστικέ καταστάσεις. Τώρα λοιπόν πάμε σε ένα σύστημα όπου ε, έχουμε με το ίδιο καθεστώς ε, τις παλές δυνάμεις και τις ανερχόμενες δυνάμεις και τις ανεπτυγμένες δυνάμεις. Νομίζω πως έχουμε ένα διάλογο λοιπόν, μια διαδικασία και όπως σας είπα δεν αναμένω από τις συναντήσεις των G20 να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα. Δεν νομίζω πως θα γίνει με αυτό τον τρόπο, αλλά σταδιακά μέσω διαλόγου είναι πάρα πολύ σημαντικό οι αναφιόμενες χώρες να αντιληφθούν πως το σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης που δημιουργήσαμε εμείς και οι Αμερικανοί ε, έχει κάποια αξία για αυτούς. Πρέπει να αναμορφωθεί αυτό το σύστημα. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν από μόνοι τους ε, πως ε, θα θέλουν να λάβουν μέρος, να ε, γίνουν μέλη με πλήρη δικαιώματα για να έχουμε μια μεταρρύθμιση. Δεν θα έχουμε επανάσταση, θα έχουμε μεταρρυθμίσεις. Και θα πρέπει να αντιληφθούν πως το σύστημα αυτό δεν θα είναι για αυτούς άδικο με τους δικούς μας ε, κανόνες, γιατί όσο σημαίνει αυτό θα έχουμε τρομερά προβλήματα. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που θα το θεωρούν ότι πράγματι συμμετέχουν και αυτοί στον ε, επανασχεδιασμό των κανόνων. Αυτό νομίζω θα ήταν φανταστικό επίτευγμα. Ευχαριστούμε κύριε Σαπίρο. Κύριε uh, Επιτρέψτε μου να σταθώ για μια ακόμη φορά στο θέμα των διαφορών ανάμεσα σε μια περίοδο κρίσης με την κανονική αντιμετώπιση του θέματος από πλευράς της ομάδας των 20 και το θέμα βέβαια που τίθεται όπως είπε ο εισηγητής είναι άλλο πράγμα το να αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα μιας κρίσης και από την άλλη να επιβάλλει μέτρα τα οποία θα αποτρέψουν την επόμενη κρίση και εδώ είναι η δυσκολία την οποία έχουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όπως είπα και στην εισαγωγή μου πως η ομάδα των 20 παραμένει ε, μια θα έλεγα ατυπική, ανεπίσημη οργάνωση κρατών και αυτό ίσως εν πολλής να είναι και ένα από τα πλεονεκτήματά της. Αυτό όμως σημαίνει ότι θέτει η κατάσταση σε πάρα πολλούς περιορισμούς ε, στο τι μπορεί να κάνει ε, μεσοπρόθεσμα η ομάδα των 20. Για μια ακόμη φορά πιστεύω λοιπόν ότι η διαρκής αξία του Δέλτα Νιτάφ θα είναι το να μπορέσει, ή θα έλεγα, να διηθήσει την ανάγκη πολιτικής παρέμβασης και σε προβλήματα τα οποία ναι μεν ε, μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν αλλά όχι με τον σωστό τρόπο. Ας αναφερθώ σαν παράδειγμα τώρα στο θέμα του κινέζικου νομίσματος και την ε, δυνατότητα υποτίμησής του. Είναι σαφές ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλές επιπτώσεις ε, σε αυτό που ονομάζουμε διεθνείς ανισορροπίες. Και γι' αυτό ακριβώς θα τολμούσα να πω ότι σαν πρόβλημα έχει δακτυλοδειχθεί από πολλούς διεθνείς οργανισμούς, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό τουλάχιστον, ακόμα και αν δούμε ποιο είναι το υπάρχον, ε, ο υπάρχον κανονισμός λειτουργίας ε, του ΔΕΛΤΑ είναι σαφές ότι θα μπορούσαν να είχαν κάνει μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε σχέση με το κινέζικο νόμισμα, κινέζικο νόμισμα στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει εφόσον δεν υπάρχει μια πολιτική βούληση εκ των έσω στην Κίνα για να γίνει κάτι τέτοιο και αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε η ομάδα των 20 ούτε το ΔΝΤ μπορεί να επηρεάσει. Συνεπώς λοιπόν προσπαθούμε να προωθήσουμε σενάρια τα οποία θα αποτρέψουν μελλοντικές κρίσεις γιατί στην ουσία αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια κάποια μετριοφροσύνη μπροστά σε τόσο σημαντικές προβληματικές καταστάσεις. Καλώς. Έχουν ζητήσει το λόγο δύο μέλη της Επιτροπής, η Ελίζα Φερέρα και η Κάθριν Στήλερ. Και μετά θα ζητήσω από τον Πίτερ Μπάξ, που είναι ο διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Υποθέσεων, για να απαντήσει. Η κυρία Φερέρα, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους προσκεκλημένους μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες τους και να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη και εδώ κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, η πρώτη ερώτηση λέει μήπως χάνουμε την κατάλληλη στιγμή την όθηση γιατί οι θεσμοί του Bretton Woods δημιουργήθηκαν αμέσως μετά την κρίση. Έχουν πια φάει τα ψωμιά τους, είναι κάπως απερχαιωμένοι και το αναγνώρισαν αυτό οι ομιλητές. Αν όμω θέλουμε μια εναλλακτική δομή, πρέπει η δομή να βγει αμέσω μετά την κρίση αυτή που βιώνουμε τώρα. Και σίγουρα γίνονται κάποιες μεταρρυθμίσεις στο ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, αλλά ακόμη δεν έχουμε μια παγκόσμια δηλωμένη πολιτική βούληση για να ξαναδημιουργήσουμε νέους ισχυρότερους θεσμούς, ούτε ο ΠΟΕ προχωρά. Οπότε οι επίσημοι θεσμοί είναι πια απειρχιωμένη, αλλά οι νέοι θεσμοί που θα αναλάβουν σημαντικά θέματα όπως το FSP και το G20 δεν είναι επίσημο, επίσημη, είναι άτυπη περισσότερο. Με αυτή την κρίση θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε τις δύο δομές, τις παλιές και τις καινούργιες ή μήπως θα χάσουμε και αυτή την ευκαιρία. Αυτή είναι μια γενικότερη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά την Προεδρία στο Φόρουμ G20, θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Γαλλικής Προεδρίας πώς ε, ε, γίνεται ένας έλεγχος ή απολογισμός μάλλον των επιτευμάτων ή των αποτελεσμάτων σε σχέση με το πρόγραμμα που έχετε. Γιατί στη διάρκεια της κρίσης τα πιο σημαντικά θέματα ήταν στο πρόγραμμα του φορουμ G20. Αλλά σταδιακά εξαφανίστηκαν ή έμειναν σε επίπεδο ομιλιών και διακηρύξεων, για τους μήκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, για το θέμα της διαχείρισης κρίσεων από τις Διεθνείς Τράπεζες, αδιαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τα προϊόντα υψηλής μόχλευσης. Είδαμε τις συμφωνίες Βασιλεία 2 και 3 αλλά είναι πολύ γενικέ και όριστε. Ε, για τους φορολογικού παραδείσους, αρχικά ο πρόεδρος Σαρκοζή είχε κάνει πολλές φιλόδοξες παρατηρήσεις και πολλά ζητήματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης και βούλης, αλλά σταδιακά επισκιάστηκαν από άλλα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο. Τι είδους monitoring κάνατε, τι παρακολούθηση ή τι εξακρίβωση αν, αυτά τα θέματα πραγματικά συνεχίζονται και υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Γιατί το κοινό βλέπει ότι το Forum G20 φτάνει σε κάποια καλή, μπαίνει σε ένα καλό δρόμο, αλλά μετά δεν υπάρχει παρακολούθηση, δεν υπάρχει συνέχεια των πρωτοβουλειών. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όντως εφαρμόζονται. Δεν βλέπουμε δεν βλέπουμε ότι τα πραγματικά σημαντικά θέματα αντιμετωπίζονται από το G20 και σε επίπεδο δράσεων. Πολλές ερωτήσεις υποβάλλεται. Θα ξαναδώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν και μετά θα ακούσουμε και τις άλλες ερωτήσεις. Με όποια σειρά θέλετε μπορείτε να λάβετε το λόγο. Ο κύριος Ζαγέ. ευχαριστώ. Για το IMS, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αναφέρουμε τόσο το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα, αλλά το Διεθνές ε, Νομισματικό και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Γιατί δεν έχουμε μόνο το σύστημα ε, ε, κειμενόμενων ισοτιμιών, γιατί υπάρχουν κειμενόμενες ισοτιμίες γιατί μερικές χώρες δεν παίζουν ε, με τους κανόνες του παιχνιδιού. Γι' αυτό μερικές ισοτιμίες είναι, μερικά νομίσματα έχουν κειμενόμενες ισοτιμίες και άλλα όχι και υπάρχουν εκεί ανισορροπίες στις, στις διάφορες ε, ισοτιμίες. Και το θέμα του ε, νομίσματος, του διεθνούς νομίσματος αποθεματικού. Νομίζω ότι προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στην ε, δημιουργία κάποιων κινήτρων και νοσμάτων για να παροτρύνουμε τις χώρες που δεν παίζουν με τους κανόνες να επανέλθουν στους κανόνες του συστήματος κειμενόμενους ε, ισοτιμιών που ήταν το σύστημα Bretton Woods. Γι' αυτό και θέλουμε αυτά τα κίνητρα να τα ενισχύσουμε και τελικά οι ασφαλιστικές δικλείδες ε, ή το δίκτυο ασφαλείας είναι να εμποδίσουμε τις χώρες να μην σωρεύουν τα αποθεματικά τους γιατί θέλουμε να έχουν επαρκή ρευστότητα σε περίοδο κρίση. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο λόγο για να συσσωρεύουν το, τα, αποθέμα, τα αποθέματά του. Είναι να μην δίνονται κίνητρα για την συσσόρευση των αποθεματικών. Είναι πολλά και περίπλοκα τα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μεταβλητότητα, το, το, της οτιμίας, το θέμα τη ρευστότητα και όλα αυτά. Για τη δεύτερη σας ερώτηση, δεν νομίζω ότι υπάρχει μια φθήνουσα πορεία, μια σταδιακή μείωση. Η πρώτη φάση θεσπίστηκε το 2008 στη Ουάσιγκτον. Εκεί κληθήκαμε να δώσουμε κάποιες άμεσες λύσεις στην κρίση και να δημιουργήσουμε ή να προσδιορίσουμε ένα πρόγραμμα προκειμένου να επιτρέψουμε σε ορισμένες οργανώσεις στο Διεθνές Ομισματικό Ταμείο και στο ε, Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να εργαστούν με βάση τη Συμφωνία της Βασιλείας. Και λάβαμε πολλές αποφάσεις για το Capital Adequacy Ratio και τους περιορισμούς. Και τελικά στα τέλη του 2010 αποφασίστηκαν, οριστικοποιήθηκαν αυτές οι αποφάσεις και θα εφαρμοστούν από τώρα. Βέβαια, δεν δόθηκε συνέχεια σε όλα τα θέματα, μερικά δεν εφαρμόστηκαν ακόμη, αλλά γι' αυτό είπαμε ότι η Γαλλική Προεδρία, η Προεδρία έβαλε στο πρόγραμμά της τη δέσμευση να εφαρμόζονται με ίσους όρους από όλες τις περιοχές του κόσμου, όλα όσα αποφασίζονται στο Συμβούλιο. Ο κύριος Μπλαβή. Για να αναφερθώ για αυτό το οποίο είπατε για την λογοδοσία, νομίζω πως στο μέλλον θα δούμε κάποια μέσα τα οποία δημιουργούνται για να μπορέσουμε και στους G20 και στο Δυντή να μπορέσουμε να έχουμε μια δεσμευσή τους. Στο μέλλον δε το Δουντού θα δημοσιεύσει μια έκθεση λογοδοσίας για να δούμε τι έχουν κάνει τα μέλη των G20 στις ε, συνόδους σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Οπότε θα δούμε τι έχει γίνει το προηγούμενο έτος. Θα έχουμε και άλλες εκθέσεις. Η έκθεση MAP που θα αξιολογήσει το οικονομικό πλαίσιο και βεβαίως θα υπάρχει και η έκθεση της βιωσιμότητας που θα αξιολογεί το πού βρίσκονται οι χώρες σε σχέση με τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Τώρα, το άλλο ζήτημα που αναφέρατε είναι περισσότερο πολιτικό ε, ζήτημα και θέλουμε να υπάρχει οπωσδήποτε κάποια όθηση σε αυτόν τον τομέα για μεταρρύθμιση του χρηματοοικονομικού τομέα. Πρέπει να πετύχουν πολλά πράγματα π.χ. στην εποπτεία και ελπίζουμε να μην χαθεί αυτή η ορμή η οποία υπάρχει. Σαπίρ. Δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα για αυτή την ορμή που αναφέρθηκε. Νομίζω πως αν δούμε όχι την παγκόσμια κατάσταση, αλλά την κατάσταση εντός της Ένωσης, μπορούμε να πούμε πως ε, εξίσου χάνεται αυτή η ορμή η οποία υπήρχε. Πριν περάσουμε στο παγκόσμιο επίπεδο με πολύ ε, ασθενέστερη διακυβέρνηση από αυτή που έχουμε στην Ευρώπη, είναι σαφές πως εάν δούμε την ε, παγκόσμια τραπεζική κρίση που είχαμε, ήδη πριν από την κρίση του δημοσίου χρέους, που βεβαίως αλληλεπιδρούν αυτές οι δύο, υπάρχουν σημαντικά διδάγματα όσον αφορά την μεταρρύθμιση, τη χρηματοοικονομική και τα θεσμικά όργανα. Βλέπω πόσα ακόμα περισσότερα έχουμε να κάνουμε και πόσο βαθιά ήταν η κρίση και πως σαφώς η απάντηση δεν ήταν ανάλογη. Και αυτά εντός της Ένωσης. Οπότε, σωστό αυτό το οποίο λέτε, πως η απάντηση και η ορμή δεν αντιστοιχούν με το μέγεθος του προβλήματος, αλλά ακόμα και εντός της Ένωσης δεν ε, καταφέρνουμε να απαντήσουμε, να αρθούμε στο επίπεδο της πρόκλησης. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, νομίζω πως πρέπει να δούμε την ε, κρίση, την παγκοσμία, στο πλαίσιο των όσων συζητάμε και που νομίζω το υπενόησαν όλοι οι ομιλητέ, δηλαδή τι αλλαγές ε, λάμβαναν χώρες στην παγκόσμια οικονομία ακόμα και πρώτη κρίση. Οπότε αντιμετωπίζουμε μια πραγματικά πολύ μεγάλη πρόκληση οικονομιών που βρίσκονται σε σχετική παρακμή η Ευρώπη και η ΕΠΑ σε σχέση με χώρες οι οποίες ε, αναφύονται ξανά θα έλεγα, όχι για πρώτη φορά, Κίνα, Ινδία και άλλες και έχουμε σοβαρή μεγάλη πρόκληση που θα υπήρχε και χωρίς την κρίση. Και η άποψή μου είναι πως η κρίση επέτεινε τα προβλήματα αυτά. Δεν τα δημιούργησε, αλλά αυτά τα προβλήματα αυτά που υπήρχαν ε, στην ε, ανακατανομή της εξουσίας και σε δημογραφικούς όρους. Θυμάστε πριν από 10-20 χρόνια όταν κοιτάγαμε τις αναπτυσσόμενες χώρες λέγαμε πως τα βασικά τους ε, προβλήματα ήταν πως ε, δεν θα αναπτυχθούν ποτέ με αυτή τη δημογραφία. Όχι. Ένα από τα προβλήματα που ε, βαραίνει τι ε, οικονομίε είναι ακριβώς το ζήτημα το δημογραφικό και τώρα που λύσαν αυτά τα προβλήματά τους το δημογραφικό είναι θετικό για αυτούς γιατί εμείς είμαστε ηλικιωμένο μέρος του κόσμου και κάποιες μέρες ξυπνάω και έχω κοιμηθεί άσχημα ε, βλέπω να πηγαίνουμε προς την Ιαπωνία Δηλαδή πλούσιοι αλλά ηλικιωμένοι με χρέος και μεγάλα προβλήματα. Και δείτε τις χώρες ε, αυτές ε, και το χρέος τους και το χρέος είπα ε, Ευρώπης και Ιαπωνίας. Και δεν είμαστε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που καταφέραμε να μειώσουμε το χρέος με γρήγορη ανάπτυξη κτλ. Δεν θα συμβεί αυτό. Δεν θα περάσουμε σε γρήγορη ανάπτυξη. Πρέπει να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν θα έχουμε υψηλή ε, ανάπτυξη και ε, πληθωρισμό. Και έχουμε γύρανση του πληθυσμού. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό με τα ωραία μας οικονομικά συστήματα και εμένα μου αρέσουν, αλλά πρέπει να μπορούμε να τα πληρώσουμε. Οπότε η κατάσταση αυτή ε, δεν, είναι, δεν είναι εύκολη. Και οι Αμερικανοί έχουν τα δικά τους προβλήματα, οι Ιάπωνες τα δικά τους. Οι βιομηχανοποιημένε χώρε έχουν τα δικά τους. Και καλά τα πάνε μέχρι Και βεβαίω έχουμε αυτές τις ε, τεκτονικές ανακατατάξεις που κάνουν την όλη κατάσταση δύσκολη. Σύντομα... Για τις δύο τελευταίες ερωτήσεις σας σχετικά με την απώλεια της ταχύτητας αυτής της όθησης την οποία είχαμε και τους στόχους τους οποίους έχει θέσει η ομάδα των 20 για μια ισχυρή και συνεχή οικονομική ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι η πρόοδος στον τομέα αυτό δεν ήταν και πολύ σημαντική. Ταυτόχρονα όμως, όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, έχει υπάρξει αρκετά σημαντική πρόοδος στο τι γίνεται ας πούμε με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα με τις νέες κεφαλουχικές απαιτήσεις των πιστοτικών ιδρυμάτων. Δεν έχουν βέβαια ολοκληρωθεί οι συμφωνίες για τα παγκόσμια λογιστικά standards, αλλά έχει υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδος. Συνεπώς δεν θα πρέπει εμείς να απορρίψουμε τα επιτεύγματα αυτά, ακόμα και αν δεν έχουμε προχωρήσει με την ταχύτητα την οποία θα επιθυμούσαμε. Σχετικά με τη δεύτερη ερώτησή σας για τη νομισματική πολιτική και το τι έχουμε πετύχει εκεί. Νομίζω ότι έχει σημασία να διακρίνουμε εδώ ανάμεσα σε αυτό το οποίο θα έλεγα ποιος είναι ο βασικός στόχος της ομάδας των 20 και από την άλλη όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία όπως είπα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις επιβαρύνουν κατά κάποιο τρόπο ε, την ατζέντα της ομάδας των 20. Ε, θυμάστε νομίζω όλοι αυτά τα οποία είχαν προτείνει οι Καναδοί όταν προείδρευαν στον τομέα ε, των μικρομεσαίων πιστοτικών παρεμβάσεων. Σαν παράδειγμα θυμάστε το νοτιοκορεατικό πλαίσιο ανάπτυξης σε σχέση με, το, με την ομάδα των 20 και το ΔΕΛΤΑ Νομίζω ότι υπάρχουν ε, ε, πολλά και τα θέματα σαν παράδειγμα των τιμών των αγαθών, των βασικών αγαθών και τα οποία υποτίθεται θα συζητηθούν αναλυτικότερα τους επόμενους μήνες. Νομίζω ότι όλα αυτά δεν θα συζητηθούν ποτέ σε βάθος και παρόλα αυτά θα επιβαρύνουν ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ομάδα των 20 και δεν θα τους αφήσουν να ασχοληθούν με τα βασικά θέματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ομιλητές μας για τα συναρπαστικά τους λόγια. Να σας ρωτήσω, το παγκόσμιο σύστημα το χρηματοοικονομικό είναι σήμερα ασφαλέστερο από ό,τι πριν την κρίση ή συνεχίζουμε όπως πριν και πώς βλέπετε το μέλλον του ευρώ. Ωραία, απαντήστε. Ε, δεν άγγει να απαντήσουν όλοι, αν θέλει κάποιος, όποιος θέλει. Um, well, very quickly on, on the <clears throat> safety of the global financial system. Well, I for certainly... Για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εγώ επενούσα την πρόοδο όσον αφορά αυτά τα οποία έκανε το σύστημα, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά θα πρέπει αυτά να τα θεωρήσουμε ως ε, έναν ελάχιστο παρονομαστή. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Και θα επιβάλλουμε τώρα υψηλότερες κεφαλαϊκές απαιτήσεις και οπωσδήποτε εγώ δεν θεωρώ για μια στιγμή πως αυτό μειώνει το θέμα εταιριών που είναι πάρα πολύ μεγάλες για να χρεοκοπήσουν. Είμαστε οριακά ασφαλέστεροι αλλά αυτό αποδεικνύει το πόσο άφρονες ήταν οι κανονισμοί της Βασιλείας 2 και οι ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά το ευρώ. Εγώ θα έβλεπα θετικά τα όσα ε, επιτέθησαν. Δεν θεωρώ πως θα συμβεί τίποτα το ανάρμοστο με το ευρώ θα παραμείνει νομίζω νόμισμα για τις 17 χώρες και θα ενταχθούν και άλλες. Αυτό δεν σημαίνει πως ε, ε, ίσως δεν θα μπορέσουμε να έχουμε μία τακτική αναδιάρθρωση χρέους, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μάλιστα, πριν περάσουμε στο δεύτερο γύρο, να ζητήσω από τον κύριο Πίτερ Μπέκ ε, Γενικό Διευθυντή της ε, Διεύθυνσης Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλύψαμε ένα ευρύτερο θέμα. Την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, το πλαίσιο για την ε, ανάπτυξη, το αριθμιστικό πλαίσιο του και τη λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και σίγουρα ένα άλλο θέμα που έχει νόημα να συζητήσουμε εδώ είναι η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν μπορώ φυσικά να καλύψω όλα τα θέματα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα επικεντρωθώ λοιπόν στα πιο ουσιώδη, κυρίως στη μεταρρύθμιση του Διεθνούς ε, Νομισματικού Συστήματος. Νομίζω ότι το μείζον πρόβλημα του συστήματος είναι ότι δεν έχει κατάλληλους μηχανισμούς προσαρμογής ε, για να αντιμετωπίσει ε, γενικές ε, ανισορροπίες. Υπάρχει ανάγκη για ε, υγιείς, βιώσιμες μακροοικονομικές πολιτικές προκειμένου να ενισχυθεί το διεθνές νομισματικό σύστημα. Το Φόρουμ G20, και εμείς δηλαδή, θα πρέπει να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις που αναλάβαμε στη Σύνοδο της Σεούλ για συναλλαγματικές ισοτιμίες και συστήματα που προσανατολίζονται προς την αγορά. Επίσης να ενισχύσουμε την γενική μακροοικονομική εποπτεία, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος του ΔΕΛΤΑ και μέσω του G20 και του ΔΕΛΤΑ ώστε να ληφθούν καλύτερα υπόψη ε, τα διεθνή spillover. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε υπέρ του έργου της Γαλλικής Προεδρίας του G20 για τις κατευθυντήριε γραμμές ό,τι αφορά τη διαχείριση των κεφαλαϊκών ροών που θα πρέπει να καλύπτουν και τις χώρες προέλευση και τις χώρες ε, ε, υποδοχής. Και βέβαια αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι μέτρα έσχατης ανάγκης γιατί η συνθήκη αποφεύγει, αποκλείει τους ελέγχους και τους περιορισμούς των κεφαλαίων. Πιστεύουμε όμως ότι από μια τέτοια απελευθέρωση θα, των κεφαλαίων θα επωφεληθεί και η παγκόσμια οικονομία. Οι οικονομίες αγορές υιοθετούν τρόπους για να προσαρτοριστούν προς την διεθνοποίηση της οικονομίας και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος να βρούμε τρόπους για περαιτέρω αύξηση της διεθνοποίησης ε, σημαντικών νομισμάτων αναδειωμένων οικονομιών και από τη στιγμή που υιοθετηθεί πρόοδος στο φόρουμ του G20 με την Γαλλική Προεδρία, θα προσπαθήσουμε να καθορίσουμε κάποια κριτήρια για να διευρύνουμε και τη σύνθεση των ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων του ΔΕΛΤΕΝΙΤΑΦ με σαφή κριτήρια προκειμένου να μπορούν και νέα νομίσματα να μπουν στο σύστημα των ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων. Τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την ενίσχυση των δικτύων ασφαλείας σε χρηματοπιστωτικά θέματα. Έχουμε διάφορες περιφερειακές νέες συμφωνίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανοίξαμε το δρόμο για καλύτερη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των περιφερειακών δικτών ασφαλείας αφενός και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αφετέρου. Επίσης τελειοποιούμε κάποιες χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις και έχουμε στενή συνεργασία και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την άποψη αυτή πιστεύουμε ότι και άλλες περιφερειακές συμφωνίες θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ευρωπαϊκών Περιφερειακών Συμφωνιών. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις. Δεν ξέρω ο κύριος Χακμαρκ θέλει το λόγο. Βεβαίως μία σκέψη, μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Καταρχήν, γιατί το G20, γιατί το φόρουμ G20. Δεν είναι απλή ερώτηση. Γιατί όμως μόνο αυτές οι χώρες είναι στο G20 και όχι οι άλλες. Γιατί άλλες σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες δεν συμμετέχουν στο G20. Γιατί δεν συμμετέχουν επίσης μερικές από τις πιο εύρυθμες οικονομίες τις οικονομίες με την καλύτερη διαχείριση. Γιατί το G20 ασχολείται με το παγκόσμιο πλαίσιο, με το γενικό πλαίσιο που θα πρέπει να ισχύει για όλους. Νομίζω υπάρχει πρόβλημα πολιτικής και δημοκρατικής νομοποίησης για το G20 όταν λέμε τι θέλουμε να επιτύχουμε σε οικονομικό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και όταν μιλούμε για ανισορροπίες, κυρίως εννοούμε τα νέα μέλη του G20. Σαν να το πρόβλημα μόνο προς τα νέα μέλη. Κύριε καθηγητά, είπατε ότι λάθος ήταν με το, τα φόρουμ G7 και G8. Αυτό. Όταν όμως συζητούμε για ενισορροπίες, κυρίως ε, εννοούμε τα πλεονάσματα. Ε, για τις ενισορροπίες όμως χρειάζονται δύο, όπως και για το ταγκό. Και μπορούμε να πιστεύουμε ότι το βασικό πρόβλημα με τις ανισορροπίες όχι, είναι όχι μόνο αυτοί που έχουν υπερβολικά καλές επιδόσεις, αλλά και αυτοί που έχουν κακές και τα πλεονάσματα δημιουργούνται και από ελλείμματα. Και αυτοί που καταναλώνουν υπερβολικά δημιουργούν τα πλεονάσματα. Και αυτό όταν το λέμε και λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανισορροπία, είναι περίεργο να περιοριζόμαστε μόνο στο G20 και δεν ε, το επεκτείνουμε σε περισσότερους γιατί αυτοί που χορεύουν το ταγκό είναι όχι μόνο αυτοί που έχουν τα μεγάλα πλεονάσματα, αλλά και αυτοί που έχουν τα μεγάλα ελλείμματα. Και βέβαια θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο για να έχουμε πραγματικά ισχυρή εφαρμογή και εποπτεία. Αν αποκλείουμε ορισμένου. Δεν υποτιμώ ή προσπαθώ να υπονομεύσω τη σημασία του Forum g G20, αλλά αν θέλουμε πραγματικά ισχυρότερο και γενικότερο παγκόσμιο αριθμιστικό πλαίσιο, γιατί να περιοριστούμε μόνο στο G20 και να μην το διαβρύνουμε σε περισσότερου ή να έχουμε περισσότερου. Γιατί όσο πιο ισχυρή και πιο εκπροσωπευτική δομή έχουμε, τόσο περισσότερα θα μπορούμε να εφαρμόσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι τα μεγάλα ελλείμματα, όπως και τα μεγάλα πλεονάσματα, σε τελική ανάλυση δημιουργούν ανισορροπίες. Θα θέσω και εγώ τώρα την ερώτησή μου, γιατί συμπληρώνει κατά κάποιο τρόπο την προηγούμενη του κυρίου Χόκμαρκ και αφορά και πάλι το G20. Αναγνωρίζουμε ότι το Φόρουμ G20 είναι μια άτυπη οργάνωση και η χρησιμότητά της έγκυται στο διάλογο που προωθεί. Είναι ένα φόρουμ διαλόγου και αυτό έχει μεγάλη αξία. Αλλά δεν υπάρχει έρχεται συνέχεια, γιατί επιλέγουμε κάποια θέματα και μετά τα παρατάμε χωρίς καμία αιτιολόγηση και περνάμε σε νέα. Και το θέμα της γραμματείας. Ακόμη και μικρές οργανώσεις έχουν τις γραμματείες τους μπορεί να, σε, είναι, να, χορηγεί, να εκχωρείται σε άλλη οργάνωση, αλλά ουσιαστικά έτσι περιοριζόμαστε μόνο σε ανακοινωθέντα τύπου με τέτοιο άτυπο, τέτοια άτυπη δομή. Ενώ για να αξίζει πραγματικά το G20 τη σπουδαιότητα που έχει, θα περίμενε κανείς κάτι περισσότερο. Έχουμε το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, που είναι μια εύρωστη οργάνωση, πολύ στεναρή, αλλά δεν τραβάει τόση προσοχή όσο το Φόρουμ G20 από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ίσως είναι πιο βαρετή κεντρική τραπεζίτες, δεν ξέρω. Επίσης έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη με πολύ καλή οργάνωση και ευρία κάλυψη θεμάτων, αλλά με αδυναμία λήψη αποφάσεων εξαιτίας της περιπλοκότητας. Οπότε διαρωτόμαστε τι θέλουμε να είμαστε στην ίδια κατάσταση με, το ΟΗΕ, με τον ΟΗΕ και τα προβλήματα που έχει να αφήσουμε το G20 ως έχει, αλλά τουλάχιστον να το ενισχύσουμε. Αλλιώς η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρασε από πολλές και διάφορες φάσεις μέσα στα χρόνια, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι για το G20, ώστε πραγματικά να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση. Για το δεύτερο σχόλιο του Γκένερ Χόκμαρτ για τον οικονομικό συντονισμό λόγω ανισορροπιών ή των ισοτιμιών. Αν πιστεύουμε ότι αυτός ο άτυπος διάλογος του G20 δεν είναι το κατάλληλο φόρουμ για να έχουμε και αποτελέσματα, μήπως θα πρέπει να διευρύνουμε την εντολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να λάβει και αυτό το σκέλος υπόψη της διορθώσης των ανισορροπιών, του μακροοικονομικού συντονισμού με τη θέσπιση δικτών κτλ. Um, Όποιος θέλει μπορεί να ξεκινήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι νιώθω ενθαρρυμένος από αυτά τα οποία είπατε και μετά από τις ε, εικονοκλαστικές της ε, αντιλήψεις που ακούστηκαν για μένα βέβαια δεν είναι παρά μια ανεπίσημη λέσχη η ομάδα των 20 ανδρών και παρότι μετέχουν και κάποιες γυναίκες είναι μια ομάδα μεγάλων χωρών που αυτό ανακηρύχθηκαν θα έλεγα η ελίτ του κόσμου αυτού. Είναι μια επιστροφή στον 19ο αιώνα όπου οι μεγάλες δυνάμεις θεωρούσαν ότι είχαν κάθε δικαίωμα όπως τη διάσκεψη του Βερολίνου να μοιράσουν τις απικίες μεταξύ τους. Δεν έχει καμία νομιμότητα, δεν έχει κανένα δημοκρατικό έλεγχο η ομάδα των 20, φυσικά είναι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και από τότε που έχουν ξεκινήσει κάνουν πάρα πολλές δηλώσεις οι οποίες ε, συνήθως δεν ακολουθούνται από πράξεις εκτός του συστήματος του Ηνωμένων Εθνών και αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα γιατί τελικά μια τέτοια μορφή διακυβέρνησης δεν θα έχει καμία μα καμία δημοκρατική νομιμοποίηση. Μάλιστα. Ιδού. G20. Ας ακούσουμε τις αντιδράσεις σας. Ξεκινήσουμε τον κύριο Ζαϊέ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στα γαλλικά. Έχω την αίσθηση ότι και οι τρεις ερωτήσεις περιστρέφονται γύρω από το κεντρικό ζήτημα, το ζήτημα της συναμοποίησης, της αποτελεσματικότητας, γιατί το Forum G20. Για το θέμα της νομοποίησης, τα 85% του παγκόσμιου ΑΕΠ, 90% με τους προσκεκλημένους, 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ε, δεν μπορείτε να μου λέτε ότι δεν υπάρχει καμία νομοποίηση. Σκεφτείτε τι αντιπροσωπεύουμε σε σχέση παγκόσμιας οικονομίας. Και όπως είπε και ο Ανδρέας Απίρ, για το G7 και G8 και η νομοποίηση για την διεθνή συνεργασία, όντως δεν υπήρχε νομοποίηση, γιατί έπρεπε να συμπεριληφθούν ε, το 99 και ήδη, όπως είπαν οι του G20, κάποιες ε, άλλες ε, συστημικές χώρες. Συστημικές χώρες όμως, όπως λέγαμε, του 99 δεν είναι κατά ανάγκη ίδιες με, με αυτές του σήμερα ή του αύριο. Η σύνθεση του G20 δεν, είναι, δεν θα παραμείνει απαράλλαχτη ή δεν μένει άθικτη. Υπάρχει ένα πρόβλημα υποεκπροσώπησης της Αφρικανικής Υπήρου. Γιατί μόνο η Νότια Αφρική επίσημα συμμετέχει στο G20. Παρόλο που προσκαλούμε, όπως είπα, και εκπροσώπους της Αφρικανικής Ένωσης, που όντως εκπροσωπούν το σύνολο των Αφρικανικών χωρών. Αλλά δεν είναι επίσημα η Αφρικανική Ένωση μέλος του G20. Όντως είναι μια λέσχη κυρίων που όμως έχουν διαφορετικές στολές, ε, κατάγονται από διαφορετικούς πολιτισμούς, έχουν διαφορετική κουλτούρα. Ε, και αυτή είναι η διαφορά σχέση με τις Βρετανικές Συλλέσιες. Και για το G20, η προστιθέμενη αξία του σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς που είναι μπορεί να έχουν περισσότερη νομοποίηση, να είναι πιο επίσημη, είναι ακριβώς η αντιδραστικότητα του φόρουμ αυτού. Η δυνατότητα αντίδραση που έχει, γιατί έπαιξε το ρόλο της σε περίοδο κρίσης οικονομικής, χρηματοπιστωτικής και δεν ξέρω αν θα έχει κάποια χρησιμότητα και σε καιρού ειρήνης. Είναι εύλογο το ερώτημα και ανοιχτό. Και σε ό,τι αφορά την Διευθύνουσα Επιτροπή ε, Οικονομικού και Χρηματοπιστικού Συντονισμού. Είχαμε το Financial Stability Board, το Συμβούλιο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας, την Επιτροπή της Βασιλείας και το θέμα για, την, ε, για τις πρώτες ύλες. Έπρεπε να δώσουμε όθηση γρήγορα για πολλά θέματα και να δώσουμε έναν οδικό χάρτη. Γι' αυτό κατάφερε να το κάνει το Forum G20 κάποια συγκεκριμένη στιγμή. Οπότε είχε ένα ιστορικό ρόλο το G20. Μπορούμε να πούμε ότι ίσως εξάντλησε εκεί το ρόλο του, αλλά θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί όπως είπα. Δεν έχει κανένα μονοπόλιο το G20 για το θέμα της γραμματείας. Ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Και το θέμα της συνέχειας. Η δική μου εμπειρία από την λειτουργία του G20 είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα συνέχειας, από τεχνική άποψη τουλάχιστον. Δηλαδή, υπάρχει μια συνέχεια των θεμάτων. Παίρνουμε τη σκητάλη από την προηγούμενη πρώτη την Κορεατική για τη διεθνή συνεργασία, το χρηματοπιστωτικό δίκτυο ασφαλεία και το καθεξής. Αλλά με όλες τις εκπεριτροπείς προεδρίας υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα γιατί κάθε Προεδρία έχει τις δικές της προτιμήσεις και προτεραιότητες για, τους συγκεκριμένους, για συγκεκριμένους λόγους, για δικούς λόγους. Και όντως κάθε Προεδρία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αποχρώσεις που ίσως ε, απομακρύνονται από μια αμυγή συνέχεια, αυστηρή συνέχεια σε σχέση με το έργο των προηγούμενων Προεδριών. Αυτά ως προς τις συγκεκριμένες επιφυλάξεις για τη συνέχεια. Τώρα για το θέμα της γραμματείας βλέποντας πώς λειτουργεί πραγματικά το G20, διαπιστώνουμε ότι έχει τεχνοκρατικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο. Έχουμε φυσικά συνεδρίαση σύνοδο, επίπεδο κρατών και κυβερνήσεων, μετά σε επίπεδο ε, επιτροπών και ε, διοικητών τράπεζας, μετά υπάρχουν διάφορε διάφορες τομεικές συνεδριάσεις, ε, γεωργικές κτλ. και τεχνικές ομάδες που δεν προεδρεύονται κατά ανάγκη από την επίσημη προεδρία του G20, αλλά μπορούν να εκχωρούνται οι προεδρίες σε άλλες χώρες. Και εκεί πάλι κινητοποιούνται συγκεκριμένες διοικήσεις. Στην πράξη είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα. Και έτσι μαθαίνουν και οι διάφορε διοικησει να συνεργάζονται μεταξύ του, όχι μόνο στα πλαίσια τη Τρόικα, αλλά και στι τεχνικέ ομάδε και υποομάδε. Και από αυτή την άποψη είναι ενδιαφέρουσα εμπειρία. Τώρα, αν θα πρέπει να προσθέσουμε και μια νέα κλίμακα με τη μορφή μια μόνιμης γραμματείας ε, στην παγκόσμια γραφειοκρατία δεν ξέρω. Και αυτό το θέμα είναι ανοιχτό πάντως. Έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας. Γι' αυτό ζητώ από τους τελευταίους ομιλητές να είναι σύντομοι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί τα θέματα αυτά έχουν ήδη τεθεί και στην παρουσίαση την οποία έκανα. Στο θέμα της αντιπροσωπευτικότητας της ομάδας των 20. Η συζήτηση αυτή που πρέπει να γίνει είναι πολιτική. Αυτό που μπορεί να δει κανείς από το Δέλτα Νιτάφ είναι ο τρόπος με τον οποίο το εκτελεστικό του συμβούλιο απέκτησε την νομιμοποίηση και παρά τα προβλήματα τα οποία έχουν συζητηθεί σε σχέση με τις ποσοστώσεις και την αντιπροσωπευτικότητα αναγνωρίζεται ο καθολικός του χαρακτήρας. Το θέμα λοιπόν είναι πολιτικό και οι αποφάσεις πρέπει να λυθούν σε πολιτικό επίπεδο. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτό. Σαπίρ να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπατε. Όπως προείπα, έχω μια θετική άποψη της ομάδας το 20, το να περάσουμε από το σημερινό σύστημα σε ένα σύστημα επιμέρους περιοχών γεωγραφικών Νομίζω ότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο δεν θα βοηθήσει πολύ και θα θέσει και πρόβλημα στην εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύντομα, όσον αφορά την εκπροσώπηση στους G20, δεν πρέπει να υποτιμούμε και την ιστορική πτυχή. Αυτό το οποίο έγινε το 2008 ήταν πως ε, κατ' ουσίαν ε, υπήρξε μια συνειδητοποίηση πως η G7-G8 δεν λειτουργούσαν, άρα χρειάζονταν μια πιο αντιπροσωπευτική ομάδα και έτυχε να επιλεγεί ε, η ομάδα των ε, G20. Κάποιες καρμαϊκές μελέτες θα σας δείξουν πως πράγματι τυχαία επιλέχθηκε ε, αυτός ο σχηματισμός αλλά βεβαίως υπάρχουν ε, κάποια πράγματα τα οποία οφείλονται σε ιστορικού λόγους. Γιατί έχουμε ακόμα πέντε μέλη μόνιμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Γιατί όταν ιδρύθηκε ο ΟΗΕ αυτοί επελέχθησαν για του γνωστούς λόγους. Όσον αφορά το άτυπο του G20, όπως ανέφερα στις αρχικές μου παρατηρήσεις, συμφωνώ πλήρως και γι' αυτό τον λόγο πιστεύω πως κύριος στόχος ε, του G20 θα πρέπει να είναι να ενδυναμώσει, όπως είπα, υπάρχοντα, υπάρχοντες οργανισμούς όπως το Βενοτού και το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας τέλος για το ζήτημα μιας ευρύτερης νομοποίησης των G20. Κοιτάξτε, δυστυχώς η νομοποίηση είναι αντιστρόφως ανάλογη με την αποτελεσματικότητα και θα μπορούσε κάποιος να πει πως ε, εντάξει καλό θα ήταν να συμμετέχουν όλοι αλλά ε, ε, εάν είχαμε κάτι σαν την Γενική Συνέλευση του ΙΕ δεν θα είχαμε παγκόσμια διακυβέρνηση οπότε είναι μια ισορροπία μεταξύ των δύο αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι όταν είναι και πάρα πολύ γύρω από το τραπέζι πάλι δεν κάνει καλό. Δηλαδή συζητάτε έναν και δικτάτορα. Αυτή είναι η ιδανική αποτελεσματικότητα λέει ο κύριος Γκέμπελς. Ήρθαμε στο τέλος αυτής της ενδιαφέρουσας συζήτησης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, δεν βλέπω, δεν βλέπω κάποιον να μας δεν λόγο. Οπωσδήποτε και ο εισηγητής και οι σκιοεισηγητές νομίζω θα τα λάβουν αυτά υπόψη τους. Ευχαριστώ λοιπόν τους προσκεκλημένους μας για τη συμμετοχή τους να υπενθυμίσω πως η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 19 Σεπτεμβρίου και θα πάει στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο το θέμα αυτό. Okay. Um, we now move on. Ωραία, περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης διαδικασίες ε, χρεοκοπίας ε, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εταιρικού Δικαίου και υπάρχει αρμοδιότητα της Επιτροπής μας για τα ζητήματα αυτά που αφορούν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αλλά Εάν ε, απομακρυνθούμε πολύ από αυτό, μετά ε, ε, θα έχουμε δυσκολίες και ίσως να μην υιοθετηθούν οι προτάσεις μας από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Μοίρασα κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και κάποιες άλλες απόψε, δεν ξέρω αν τις έχετε όλοι λάβει. Ε, λαμβάνοντα υπόψη ε, κάποιες απόψεις των πρασίνων. Το απλούστερο που μπορώ να κάνω είναι νομίζω να σας πω το τι προτείνω στις συμβαστικές τροπολογίες. Γιατί οι περισσότερες νομίζω ήταν θετικές. Πρώτη τροπολογία που προτείνω είναι στην παράγραφο 1 όπου λέω φρονεί ότι οι διασυνοριακές διαθήκες σε ζωή πρέπει να είναι νομικά εκτελεστές ε, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ε, συστημική σημασία, ακόμα και αν δεν είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης των κρίσεων, λαμβάνοντας υπόψη, όπως σας είπα, τροπολογία των σοσιαλδημοκρατών πιθανόν να μην ε, ικανοποιείται από το δεύτερο μέρος η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αλλά νομίζω πως το πρώτο μισό θα μπορέσουμε να του αναγκάσουμε να το δεχτούν. Προτείνω επίση μια δεύτερη συμβαστική τροπολογία που θα λέει τρο... τονίζει πως η διασυνοριακή χρακοπία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού εταιρικού Δικαίου θα πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός ευρωπαϊκού γενικότερου πλαισίου διαχείρισης με ελάχιστη κοινή δέσμη κανόνων και τελικά ένα κοινωνικό σύστημα για, επιχει... για επίλυση με κρίσεων. Γιατί ε, να πούμε πως ε, το καθώς αυτό της αφαιρεγγαιότητας βεβαίως είναι μέρος μόνο της όλης της ε, διαδικασίας των όσων κάνουμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο διαχείριση των κρίσεων. Μετά στην παράγραφα 2. Φρονεί ότι οι συνεργικές διαθήκες ζωής πρέπει να προβλέπουν ε, ξεχωριστές διατάξεις για βιώσιμες μονάδες που παρέχουν απαραίτητες ε, υπηρεσίες όπως συστήματα πληρωμών. Είναι σαφές νομίζω για το ήθελα αυτό. Και προτείνω ε, να προσθέσουμε κάποιες διατυπώσεις που είχαν για να συμπεριλαμβάνει διατάξεις για διαχωρισμό διασυνοριακών ομίλων σε βιώσιμες ομάδες. Μα, κυρία Πρόεδρε, οι διερμηνείς μας λένε πως δεν έχουν το κείμενο από το οποίο εσείς διαβάζετε τις ε, τροπολογίες. Ε, δεν ξέρω αν μπορείτε να τους το δώσετε. Ή αλλιώς, ε, γιατί βλέπετε, οι δυο μας και ένας τρίτος είναι σε αυτή την ωραία αίθουσα, εδώ είναι. Λοιπόν, μπορείτε να μας παρουσιάσετε συνοπτικά τις απόψεις σας. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία, θα είμαι σύντομη, τότε μην τα διαβάσω όλα αυτά. Αυτό το οποίο έκανα είναι ότι συγχώνευσα τις τροπολογίες η βασική διαφορά νομίζω σε σχέση με αυτά τα οποία είχατε εσείς είναι πως το περιορίσατε λίγο στις τράπεζες, εγώ προσπάθησα να το κάνω κάπως ευρύτερο πέρα από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, νομίζω στην οπολογία 7. Και το άλλο βασικό τμήμα της διαφοράς που είναι στο τελευταίο πιο πρόσφατο κείμενο που απέστειλα είναι κάποιες διατυπώσεις των πρασίνων που είχε αναφέρει ο Σβέν που βασίζονταν στο να συμπεριλάβουμε ομίλους και νομίζω πως ήταν λογικό να συμπεριλάβουμε και τους ομίλους εφόσον είναι στην αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Οπότε όταν μιλάμε για διαχωρισμό νομίζω είναι σημαντικό ε, για τις περιπτώσεις ε, ομίλων ε, και για τον απομισθούν και οι μέτοχοι κάποιο βάρος στις περιπτώσεις αυτές και μπορούσαμε να έχουμε αντίστροφα τεστ κοπόσεως στην περίπτωση των ομίλων, κάτι το οποίο νομίζω γίνεται ήδη στο πλαίσιο των τραπεζών. Αυτά ήταν τα επιπλέον κομμάτια που πρότεινα να, να μπουν ως συμβιβασμοί με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ αν τους έχετε δει και είστε διατεθειμένοι να τους δεχτείτε. Κανένα πρόβλημα. Ε, δεν νομίζω πως υπήρχε καμία ασυμβίβαστη διαφορά. Ε, θα περιοριστώ σε αυτά. Ε, Ζαν Πολ, θέλεις το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, μετά αυτό το ενθουσιώδες πλήθος που παρακολουθεί ε, αυτή την έκθεση, ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι και εγώ τις θέσεις σας και δεν έχω άλλες παρατηρήσεις για το κείμενο. Σας ευχαριστώ θερμά για, το έργο σας και την, ε, και την γνωμοδότηση. Ο Σαΐντ. Σαΐντ, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Ε, μπορεί να μας παρακολουθούν από το ίντερνετ και το web stream. Εν πάση εδώ πέρα δεν είναι πάρα πολύ, αλλά συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπατε. Είναι πάρα πολύ καλή έκθεση. Έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες, ε, επί των οποίων υποβάλλατε κάποιες συμβαστικές προτάσεις και εγώ μπορώ να τις στηρίξω, τις προτάσεις σας. Πράγματι, Βεβαίως ε, υπήρχε ένας περιορισμός στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θεωρώ ότι είναι θετικό να το δούμε ευρύτερα το ζήτημα. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε πως είναι πολύ σημαντικό ο τομέας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εκεί πέρα χρειάζονται ε, κανόνες για να εναρμονιστεί το ζήτημα της ε, αφαιρεγγιότητας. Και πράγματι αυτές οι διαθήκες εν ζωή είναι πολύ σημαντικό βήμα. Αυτά πράγματι είναι πολύ θετική η πρόταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, το ζουμί το πιάσατε. Είναι εκεί που δημιουργήσαμε δηλαδή εργαλεία στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών ενδρυμάτων. Δεν ήθελα να γίνει κάτι στο πλαίσιο της αφαιρεγγιότητας για να αφαιρεθούν αυτά τα εργαλεία. Πρέπει να τα επεκτείνουμε να υπάρχει μια ακόμη μεγαλύτερη διασυνοριακή διάσταση, όπου αυτό είναι δυνατόν. Εάν δείτε δε λεπτομερώς τις συμβαστικές προτάσεις, ε, υπάρχουν... Ε, αν σκεφτείτε και κάποια άλλη ιδέα, ευχαριστώ να τεχτώ. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε 12 Ιουλίου, οπότε υπάρχει λίγος χρόνος για έτσι, κάποιες αλλαγές ή και για να εισαχθεί κάτι άλλο που εσείς θεωρείτε σημαντικό. Η ψηφοφορία στην ε, κατά κύριο λόγο αρμόδια επιτροπή είναι στις 9 Σεπτεμβρίου, οπότε υπάρχει χρόνος. Και νομίζω πως μπορούμε τώρα να περάσουμε στα διάφορα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, οπότε λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ. We meet again in Strasbourg on the 4th of July.